Euh, Καλημέρα σας. Προτείνω να ξεκινήσουμε την συνεδρίαση. Θα έχετε δει ότι έχουμε αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στην κινητικότητα πάνω από όλα σήμερα. Απλώς ε, μια επισήμανση Ίσως κάποιοι αύριο να έχουν δυσκολία να φτάσουν στο κοινοβούλιο γιατί αναμένεται αύριο στο Βέλγιο μια απεργιακή κινητοποίηση στο δημόσιο τομέα και στις δημόσιες ε, στις σημασικές μεταφορές, οπότε μπορεί η τηλεφορία και τα μετρό να μας δημιουργήσουν κάποιες δυσκολίες. Θα αρχίσουμε στις 9.30 λοιπόν και αυτό πάλι με την ελπίδα ότι θα έχουμε την απαρτία ώστε να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες και να επεξεργαστούμε τα διάφορα θέματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Ε, ενημερωτικά τώρα, οι Ανιές Ιόγκερης είναι εδώ μπορούμε να δούμε τα θέματα για την ε, οδηγία, για την ε, απόσπαση ενιές. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και διαρωτώ εάν ε, το απεργιακό κίνημα του Βελγίου συντονίζει τις δράσεις του, τι με τις δικές μας συνεδριάσεις. Ελπίζω ότι θα είναι μόνο σύμπτωση. Στην απόσπαση Έχουμε τον 7ο τριμερή διάλογο στο πρόγραμμά μας τη Δετάρτη και νομίζω μπορούμε να πούμε εν γέννη ότι είμαστε σε συμφωνία σε σχέση με τις συλλογικέ συμβάσεις σε σχέση με τις αμοιβέ. Έχουμε συζητήσει τις αμοιβέ και πιστεύω λίγο πολύ το έχουμε ολοκληρώσει. Πέντε θέματα ωστόσο παραμένουν. στο τραπέζι των συζητήσεων ε, που μας διχάζουν εμάς με το Συμβούλιο και εν μέρει και την Επιτροπή. Καταρχάς το, η διάρκεια της απόσπασης 24 μήνες συν παράταση για το Κοινοβούλιο ενώ το Συμβούλιο λέει 12 συν 6 και η Επιτροπή υποστήριζε τους 24 μήνες. Υπάρχει ένα θέμα επίσης σε σχέση με τον τομέα των μεταφορών, που βεβαίως έχει τη σημασία του εξιστής μας εδώ, στην Επιτροπή μας. Γιατί λέμε στη γνωμοδότησή μας ότι οι μεταφορές πρέπει να είναι κομμάτι της νέας οδηγίας έχει κάνει μια προφορική τροπολογία του Συμβούλου, μια συμφωνία προφορική. Ένα τρίτο θέμα είναι η νομική βάση. Ένα άλλο θέμα είναι η υπεργολαβία. Και έχουμε και θέμα σε σχέση με την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή όπου το Συμβούλιο αντί των συνήθων δύο ετών ε, επεξεργάζεται λύσεις τριών και τεσσάρων ετών για την εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο. Μεταφορά και εφαρμογή. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που μας διχάζουν ακόμη. Πρέπει βεβαίως να καταλήξουμε και σε διαφορές άλλες θέσεις. Πρέπει να δούμε τις αιτιολογικές σκέψεις. Πάντως και η Επιτροπή και το Συμβούλιο φαίνεται να ενδιαφέρονται για μια γενική συμφωνία για τις επόμενες εβδομάδες αισθάνομαι όλο και μεγαλύτερες τις πιέσεις που μου ασκούνται. Για... Αλλά βέβαια προσπαθώ και εγώ να εξασφαλίσω μια καλή και ισορροπημένη συμφωνία. Περισσότερα μετά την Τετάρτη. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ, Όνιες. Έχετε άλλωστε συνάντηση με τους Σκιώδη σήμερα, έτσι, μετά τη συνεδρίαση. Στις 28 στο Συμβούλιο για τη διερμηνία. Είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες πλην της φινλανδικής, της βουλγαρικής και της κροατικής γλώσσας. Ζητώ συγγνώμη επίσης εκ μέρου της Μαρίτα τη Προέδρου μας που απουσιάζει, θα έρθει αργότερα, έχει μια μικρή καθυστέρηση στο αεροπλάνο τη. Αναλαμβάνω λοιπόν εγώ να προεδρεύσω μέχρι ότου φτάσει και η Μαρίτα. Και ξεκινούμε με το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Έκθεση για τις απαιτήσει εφαρμογή και ειδικοί κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών. Με τη Μαρτίνα Τλαμπάιωβα, η Παρακαλώ. Σας ε, ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλους σας. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τις συναδέλφους ε, για τις 367 τροπολογίες που κατατέθηκαν ε, σε αυτή τη γνωμοδότηση. Το θέμα της απόσπασης των οδηγών είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή και οτιδήποτε πείτε έχει μεγάλη σημασία. Ανέλησα λοιπόν όλες τις ε, τροπολογίες και διαπίστωσα ότι υπάρχουν ε, και κάποιες σημαντικές απόψεις που έχουν ε, κατατεθεί. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να δούμε και πώς θα μπορούμε να είμαστε και δημιουργικοί στο θέμα των συμβασμών. Να σε εξηγήσω λιγάκι τη στάση μου απέναντι σε αυτό το θέμα και τι πρέπει να κάνουμε ως και οδησηγητές. Το θέμα είναι να βρούμε μια λογική, τεχνικά εφικτή λύση, να προσπαθήσουμε κατά κάποιον τρόπο να ξεπεράσουμε τις πολιτικές διαφορές. Εγώ θέλω να υπάρχουν κανόνες ε, που να μπορούν να εφαρμοστούν και που θα δώσουν τη δυνατότητα στους ε, μεταφορείς να εφαρμόζουν αυτούς τους ε, κανόνες ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και κοινωνικές εγγυήσεις και εξασφαλίσεις για τους οδηγούς. Επ' αυτού πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε να βρούμε μια λύση για να υπάρχει ισορροπία. Στην Επιτροπή μας οι κανόνες που αφορά την ε, αμοιβή των εργαζομένων προκύπτουν από τη γενικότερη οδηγία περί απόσπαση των εργαζομένων. Και όπως ακούσατε ήδη, αυτή η γενική είναι υπό αναθεώρηση. Συζητάμε ε, νέους κανόνες ε, όπως θέμα αμοιβή, υπεργολαβίες. Τα αναθεωρούμε όλα. Άρα δηλαδή και όσον αφορά τη ρήτρα περί μεταφορών που θα μπει στη γενική οδηγία, εκεί θα υπάρχει δική εφαρμογή του Lex Specialis. Για το λόγο αυτό, στη δική μου, στο δικό μου το σχέδιο γνωμοδότηση έχω εξαιρέσει τις διεθνείς μεταφορές και την, ε, το διαμετακομιστικό εμπόριο, γιατί είναι αδύνατον οι νέε διατάξεις για την ε, απόσπαση των εργαζομένων να εφαρμόζονται σε ένα τομέα με τόσο μεγάλη κινητικότητα όπως είναι οι μεταφορές. Αν μπορεί κάποιος ε, να μου εξηγήσει το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτούς τους κανόνες σε κάποιον που αλλάζει χώρα ανά δύο-τρεις ώρες, ε, πώς ε, μπορούμε να επιτρέπουμε το καμποτάζ ή οτιδήποτε άλλο. Αν μπορούσε να μου το εξηγήσει, ίσως να άλλαζα γνώμη. Αλλά δεν νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν στην πράξη. Κατά, την, κατά τα άλλα, όσον αφορά τα προβλήματα που ανέφεραν ορισμένα κράτη-μέλη, εγώ το καμποτάζ το περιλαμβάνω από την πρώτη μέρα της απόσπασης, ε, βέβαια με μια πιο σταθερή μορφή. Υπάρχουν διάφορες ε, τροπολογίες ε, που εκφράζει την άποψή σας, οφείλουμε να βρούμε μία λύση. Lex specialis. Ε, είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η μορφή κανόνα. Το θέμα πρέπει να ληφθεί με την μη τυπική εφαρμογή των κανόνων και νομίζω ότι αυτό τρέχει εδώ και κάποια χρόνια στα κράτη-μέλη. Βλέποντας αυτά που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοί μου και την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με τους και ηγητές, πραγματικά πιστεύω ότι οφείλουμε να βρούμε ένα κοινό παρανομαστή και θα τον βρούμε τελικά. Οφείλουμε να δείξουμε στην κοινή γνώμη ότι ως κοινοβούλιο μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε εφικτές λύσεις οι οποίες ξεπερνάνε το πολιτικό στενό πλαίσιο. Αυτή είναι η γενική μου τοποθέτηση και με μεγάλη χαρά να ακούσω τις παρατηρήσεις και μετά στο τέλος θα μου επιτρέψετε να κάνω έτσι και μια συμπερασματική παρέμβαση. Εκ μέρους του ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το ότι η συνάδελφός μας ε, δεν μπορεί να είναι παρούσα. Έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα όπως και η κυρία Πρόεδρος. Δηλαδή έχει καθυστερήσει η πτήση τους και αυτός είναι ο μόνος λόγος ε, που την εμπόδισε να είναι στην ώρα της. Με παρεκάλεσε λοιπόν να παρουσιάσω τη θέση της που είχε προετοιμάσει για τις σημερινή συνεδρίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο τομέας των μεταφορών είναι ένας ιδιαίτερος τομέας που χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα των εργαζομένων. Γι' αυτό, ειδικά εδώ, στον τομέα αυτό, χρειαζόμαστε κανόνες που να είναι σαφείς, ε, κατανοητοί, εφικτοί και να μπορούν και να ελέγχονται. Χρειαζόμαστε κανόνες ε, που θα επιτρέπουν τη λειτουργία αυτού του τομέα, ε, λειτουργία προσαρμοσμένη και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ασχολούμαι πολλά χρόνια με την απόσπαση και γνωρίζω πολύ καλά πόσο περίπλοκο είναι το θέμα. Πλήρη εφαρμογή των κανόνων ε, αυτό μπορεί να γίνει σε άλλους τομείς, ε, ας πούμε στον τομέα των κατασκευών, αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η εφαρμογή στον τομέα των μεταφορών. Οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και δεν υπάρχει πλειοψηφία για μία ενιαία λύση. Γι' αυτό χαίρομαι που όλοι οι σκιώδεις εισηγητές ε, προτιμοποιήθηκαν το θέμα να το αντιμετωπίσουν αντικειμενικά και να μην κολλήσουν σε μικροπολιτικές επιφυλάξεις. Κατά τις επόμενες εβδομάδες. Πρέπει να καταθέσουμε πρόταση για τις διεθνείς μεταφορές, για το καμποτάζ. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία ε, συμβαστική πρόταση σχετικά με τους κανόνες περί απόσπασης. Άλλο θέμα σημαντικό είναι ο έλεγχος και η εφαρμογή των κανόνων. Χαίρομαι που έχουν κατατεθεί καλές τροπολογίες από αυτού. Από ό,τι φαίνεται συμφωνούμε ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επεξεργαστεί ένα συγκεκριμένο έγγραφο που να οδηγήσει σε μείωση του διοικητικού φορτίου. Εμείς ως ΕΛΚ θα ταχτούμε υπέρ των αυστηρών ελέγχων και της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ο έλεγχος να γίνεται ηλεκτρονικά. Πολλοί βουλευτές έχουν προτείνει αυτό το σύστημα να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του ΕΜΗ, του συστήματος περί κοινή αγορά. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν πολύ εύκολα να καταγράφονται και να επικαιροποιούνται τα δεδομένα. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε μια κοινή πρόταση που να αφορά στις αμοιβέ και στις συμβάσεις. Ε, τα έγγραφα αυτά πρέπει να ελέγχονται στον, στην έδρα της εταιρείας γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο καθοδόν και νομίζω αυτό το προτείνουν και πολλοί άλλοι βουλευτές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εφαρμοστική οδηγία για την απόσπαση περιλαμβάνει σαφείς διατάξεις για το πώς πρέπει να γίνεται ο έλεγχος χρησιμοποιώντας κυρίως το σύστημα Ε, Η επεξεργασία καλών δεδομένων απαιτεί βέβαια υπευθυνότητα εκ μέρους μας όπως και ανοιχτό πνεύμα. Το γεγονός ότι ως προς την επεξεργασία της οδηγίας περί απόσπασης δεν υπάρχει συμφωνία αυτό μας απασχολεί. Συνεχίζονται οι τριμερείς διάλογοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι νέοι κανόνες θα αφορούν τον τομέα των μεταφορών. Γι' αυτό θα πρέπει με την ησυχία μας να ελέγξουμε τους κανόνες για την απόσπαση των εργαζομένων, να ελέγξουμε κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα. Ορισμένες τροπολογίες καθιστούν σαφές ότι στον τομέα των μεταφορών όπου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόζονται οι κανόνες για την μακρο μακροπρόθεσμη απόσπαση. Δύσκολο και για τις ε, συλλογικέ συμβάσεις που δεν είναι γενικής φύσεως. Γιατί με τον τρόπο αυτό επιβαρύνονται υπερβολικά οι μεταφορικές εταιρείε, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται και ουσιαστικά ωφέλη για τους εργαζόμενους. Ελπίζω οι συναδελφοί να λάβουν υπόψη τους την κατάσταση. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ μεγάλη. Ε, έχουμε μπροστά μας ε, πολλές ευθύνε, πρέπει να είμαστε συνετοί. Πάρα πολλοί συνάδελφοι επισημαίνουν και το πρόβλημα των των ε, εταιριών γραμματοκιβώτιο ε, με κανονικούς όμως ε, εργαζόμενους υπάρχει και το πρόβλημα των φορτηγών κάτω από 3,5 τόνους και τους ήμι απασχολούμενους. Αυτά είχα να σας πω και σε σχέση με την οδηγία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρέγνερ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θυμίσω λίγο το σημείο αφετηρίας. Μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπινα όντα τα οποία δουλεύουν σκληρά. Και ε, πρόκειται για ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά όταν είναι διέλευση, όταν είναι διεθνείς μεταφορές, όταν είναι καμποτάζ. Πάντοτε λοιπόν πρόκειται για τις ε, συνθήκες εργασίας και την υγεία των ανθρώπων που κάθονται πίσω από το τιμόνι. Τώρα να βρούμε πάρα πολύ στεριά κριτήρια ε, για τους ελέγχους και να λέμε είναι καμποτάζ, είναι κάτι άλλο. Πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους αυτούς πώς είναι ώρα κάθονται στο φορτηγό, μπορούν να κοιμηθούν καλά, αξιοπρεπώς, περί αυτού πρόκειται. Δεν ε, είναι μόνο θέμα εσωτερικής αγοράς, ε, κυκλοφορίας ε, και ολόκληρης κινητικότητας αυτό του τομέα. Πρόκειται για τους ανθρώπους αυτούς που κάθονται εκεί μέσα στο φορτηγό. Και γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ σήμερα στην Επιτροπή και αποφασίσαμε ότι όταν μιλάμε για την απόσπαση πρέπει να μιλούμε για όλους όσους βρίσκονται υπό απόσπαση γιατί όλοι χρειάζονται κάποιο είδους προστασία. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στη συνάντηση σκιωδών εισηγητών που είχαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ ε, την Μαρτίνα Τλαμπάγιοβα, την εισηγήτριά μα γιατί είχα την εντύπωση, προφανώς εδώ έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις ε, μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων, ε, Νομίζω όμως ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το επικοδομητικό πνεύμα ως ε, συνάδελφοι που θέλουν να καταλήξουν σε ένα ε, συμβιβασμό και να μην μιλούμε απλώς για ε, αδιάλακτες τοποθετήσεις σε σχέση με τους ανθρώπους αυτούς. Την επόμενη φορά λοιπόν να το έχουμε αυτό υπόψη μας όταν θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα συμβιβασμό. Κάτι ακόμη οι συμβιβασμοί είναι, καλό είναι να εξευρεθούν, να υπάρξει ένα κείμενο που να επιτρέπει σε όποιον ε, οδηγεί ένα φορτηγό να έχει ένα, αυτό, ένα πλεονέκτημα με αυτή την διπλή νομική βάση. Εγώ όχι μόνο είμαι υπέρ του συμβιβασμού, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε πιο αυστηρούς τους ελέγχους και να επιβάλλονται σωστά. Υπάρχουν όμως πολλά νομικά, ε, πολλά παραθυράκια στην ομοθεσία. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της οδηγίας επιβολής, είναι το ζήτημα της ίδιας απόστασης, της απόσπασης ε, που πρέπει να εξετάσουμε. Και επίσης ε, υπάρχει ένα παζάρι για τις ημερομηνίες στο Συμβούλιο, το διαπιστώνουμε τι κάνουμε τώρα, προστατεύουμε πράγματι αυτούς τους ανθρώπους που οδηγούν τα φορτηγά με αυτές τις συζητήσει. Η λύση που θα βρούμε η τελική μας λύση πρέπει να είναι μια λύση που θα προστατεύει καλύτερα τους οδηγούς αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν είναι κανείς εδώ από την ECR. Οπότε τώρα περνάμε στους πρασίνους. Στην ΚΟΕ, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Πατρίκ που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τα εισαγωγικά της σχόλια, όπως επίσης και για τις προτάσεις της. Αυτό που μας απασχολεί προφανώς περισσότερο είναι η προστασία των εργαζομένων να μείβονται σωστά και οι συνθήκες εργασίες τους να είναι καλές. Ε, Γι' αυτό είχαμε υποβάλει και τις σχετικές τροπολογίες. Θέλουμε το πεδίο εφαρμογής να είναι αρκετά ευρύ. Γιατί τι πρέπει να ρυθμίσουμε, πρέπει οι συνθήκες να είναι καλές στον τομέα των οδικών μεταφορών. Πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν περισσότερες δυνατότητες διενέργειας ελέγχων και προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται οι προτάσεις τροπολογιών μας. Γι' αυτό πρέπει όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι να προστατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο και τα κράτη-μέλη να μπορούν να κάνουν σωστούς ελέγχους και να εφαρμόζονται τα μέτρα σωστά. Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους οδηγούς και ο κανόνας, οι κανόνες επί απόσπασης ε, είναι νέο, νέοι κανόνες ε, οι οποίοι βρίσκουν μια ισορροπία μεταξύ του ανταγωνισμού και της προστασίας των εργαζομένων. Αυτό ακριβώς είναι η λογική πίσω από τα νέα αυτά κανόνα, αυτοί αυτοί κανόνες. Κυρία Ρέν Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τη Ματίνα για το σχέδιο. Χάρη και στους άλλους σκιώδες ηγητές έχουμε ένα καλό σημείο αφιτερίας που εκδηλώθηκε ήδη στην προηγούμενη συνεδρία των σκιωδών. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα γεγονός της προηγούμενης εβδομάδας. Ένας Τσέχος οδηγός λεωφορείου που εργαζόταν για την Deutsche Post AG της Γερμανίας ελέγχθηκε και από τις πληροφορίες που έλαβε κατά τη διάρκεια του ελέγχου ενημερώθηκε ότι ε, θα έπρεπε να παίρνει τον ελάχιστο μισθό το γερμανικό ενώ τον πλήρωνε το 1 τρίτο αυτού του ποσού και έχει κάνει μήνυση, έχει κάνει αγωγή. Έχει κάνει αγωγή λοιπόν και τελικά η Deutsche Post AG αποφάσισε να του ε, καταβάλει τη διαφορά, τα 2 τρίτα δηλαδή, αναδρομικά γιατί καθώς οδηγούσε φορτηγό στη Γερμανία έπρεπε να αμείβεται με το γερμανικό ελάχιστο μισθό. Αυτό χωρίς απόφαση δικαστική εντωμεταξύ διότι επήλθε συμφωνία αλλά μας δείχνει ότι κάθε πλευρά, κάθε εμπλεκόμενη πλευρά χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια. Είναι πολλά τα, πολλά τα κενά του νόμου και τα παραθυράκια που οδηγούν στο να μην υπάρχει ενιαία λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθήκον μας είναι και να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή και υλοποίηση της νομοθεσίας και τους ελέγχους στην κάθε χώρα. Πρέπει επίση να πω με πάσα ειλικρίνη ότι διαβάζοντα τι προτάσει τη Επιτροπή δεν διαπιστώνω ότι θα εξασφαλίσουν περισσότερη διαφάνεια τόσο για του εργαζομένου όσο και για τι μικρομεσαίε ή τι μικρότερε επιχειρήσει που μπορεί να μην έχουν ε, εκτεταμένε ομάδε νομικών ε, παραστατών. Ε, αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερο χάο. Γιατί δεν υπάρχει σαφή αντίληψη. Ο καρόνα για τι τρει ημέρε δεν νομίζω ότι βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην υλοποίηση αυτών των κανόνων και τη βελτίωση εκ τούτου των συνθήκων εργασίας των οδηγών και γι' αυτό για μένα ε, σαφής ως προς την εφαρμογή τους κανόνες είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορούμε να επιδιώξουμε και όπως είπαν και οι συνάδελφοι σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς δηλαδή θα πρέπει να ενημερώνονται για τη νομοθεσία και, τη, και να την υλοποιούν σωστά. Αυτό που βλέπουμε και στον τριμερή διάλογο για την απόσπαση εργαζομένων είναι ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια μέσω ενός ε, εθνικού ενιαίου εθνικού ιστοτόπου, πολύ σημαντικού και για τις μεταφορές και επίσης αυτό εάν πρόκειται για την ε, αξιολόγηση του τι συμβαίνει στην κάθε χώρα, στην ε, αγορά των μεταφορών ε, νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει ιδιαίτερα το σύστημα του ταχογράφου. Και κάτι ακόμη, μπορεί να μην έχουμε μεγάλες διαφωνίες στο θέμα αυτό και χαίρομαι που και άλλοι συναδελφοί ανέφεραν πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά όλα τα μέτρα ελέγχου, αυτά τα μέτρα τα οποία απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η, η επιβεβαίωση της στήριξης των κανόνων, είναι ότι πιο σημαντικό, γιατί πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση να υφίσταται νομοθεσία, να ισχύουν κανόνες, αλλά να μην τηρούνται, να μην υλοποιούνται. Αυτό λοιπόν πρέπει να το επισημάνουμε ότι θα υπάρχει και ένας κατάλογος ε, ενδεικτικός μέτρων ελέγχου. Ευχαριστώ. Η FTD υπάρχει κανείς εδώ. Κύριος Ντομίνικ Μαχτάν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μαρτίνα. Ιδιαίτερα εκτιμώ αυτό το τεράστιο έργο, αλλά και τις, ε, τα προσωπικά χαρίσματα, την ευγένεια και τη διάθεση συνεργασίας. Αρχικά είχαμε αντιταχθεί στο να αποσπαστεί από την ε, οδηγία για, την, ε, για τους αποσπασμένους εργαζόμενους στο θέμα των μεταφορών. Γιατί υπάρχει η ε, διαμετακόμιση, το καμποτάζ, το οποίο οδηγεί σε διαφορετική μεταχείριση αναλόγως ως προς τους εθνικούς μεταφορείς και εργαζομένους. Εγώ μεγάλος και δεν διστάζω να πω πρώτα οι Γάλλοι. 28.000 θέσει εργασία έχουν καταργηθεί τα τελευταία χρόνια, σε 10 χρόνια μέσα. Και σε 10 μέσα χρόνια έχουν ε, εξαφανιστεί ε, το 1 τρίτο των επιχειρήσεων των μεταφορών σε εθνικό επίπεδο. Ενώ η λύση είναι πολύ απλή. Αρκεί να απαγορευτεί η διαμετακόμιση, το καμποτάζ. Και όπως είπε και η προλαλή σας, ε, Ας μην αρχίσουμε αυτές τις, αυτό το παιχνίδι ε, της ε, επιλεκτικής ανάγνωσης τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, πέντε μέρες, ένα σύστημα δηλαδή μέσα στο οποίο εξασφαλίζεται η εκμετάλλευση του εργαζομένου, αρκεί να απαγορευτεί η διαμετακόμιση. Μια επιχείρηση έχει να μεταφέρει από το κράτος Α στο κράτος Β της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπορεύματα. Ένας διεθνής μεταφορέας μπορεί να κρατάει την αγορά να προβαίνει στην παράδοση, στη μεταφορά και παράδοση και αν είναι ικανός μπορεί και να επιτύχει να ξαναφορτώσει για να επιστρέψει ή για να πάει να παραδώσει σε άλλο κράτος μέλος, να μην γυρνάει άδειος δηλαδή. Και έτσι, Μαρτίνα, αν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε αυτό, με βέβαιος ότι θα βρούμε μια απλή λύση. Ως προς τον ταχογράφο. Τέλεια, τα καταφέραμε πάλι. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι απαραίτητο να ελέγχεται ο χρόνος οδήγησης, ο χρόνος που είναι κανείς στο δρόμο, ο χρόνος ανάπαυσης, ο χρόνος επανόδου στην εστία του καθενός. Μα σας υπενθυμίζω ότι υπάρχουν και περιβαλλοντικοί κανόνες και υγειονομικοί κανόνες και κανόνες για την ε, ευημερία των ζώων κανόνες ασφαλείας που παραγνωρίζονται απολύτως. Τους ξεχνάτε. Και βεβαίως πρέπει να προστατευτεί ο οδηγός. Άνθρωπος είναι, το πάτε κι εσείς. Αλλά όλα τα άλλα. Το μεταφερόμενο προϊόν. Η χρήση των υποδομών μας, των οδικών υποδομών. βλέπουμε ατυχήματα δεξιά και αριστερά. Γιατί είναι ακριβώς αυτοκινητόδρομος, οπότε θα προτιμήσουμε τον εθνικό δρόμο. Και δεν πληρώνουμε σε τίποτα την ε, φθορά των υποδομών της χώρας στην οποία διανύουμε, διασχίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Αυτή η μεταφορή, η low cost μεταφορής, θα πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν στην ε, χώρο ταξίας, στην αποκατάσταση των υποδομών. Φανταστείτε, μια χώρα όπως η Ελβετία, η οποία δεν έχει διόδια για τον Ελβετό στους δρόμους της, αλλά για το μη Ελβετό επιβάλλει τη δινιέτα, η οποία σημαίνει ότι και μάλιστα θα μιλήσω για τη χώρα μου, τη Γαλλία, που την προτιμώ όπως και να είναι, θα πρέπει να καταβάλει κανείς το μερίδιο, το τίμημα που του αναλογεί. Μαρτίνα, αυτό είναι και το αντικείμενο των 29 τροπολογιών μου. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Μια δήλωση μόνο για το σύνολο των τριών κειμένων που θα μας απασχολήσουν το ένα μετά το άλλο, γιατί αποτελούν ένα σύνολο. Καταρχάς ευχαριστώ τους τρεις εισηγητές, τη Μαρτίνα Γατλαμπάζοβα, τον φίλο και, Μπαχ και την κυρία Λόπες Φοντανιέ, τη φίλη, για τη δουλειά που έχουν κάνει στα τρία κείμενα. Αυτά προσωπικός αλλά και εξ ονόματος των Γάλλων πολιτών και ως μέλος της Επιτροπής. Λυπούμε λοιπόν, ωστόσο που κάποιες από τις, φιλοδο... δεν είναι αρκετά φιλόδοξε, από ό,τι βλέπω εγώ και δεν είναι προσαρμοσμένες στις πραγματικέ συνθήκε που επικρατούν στις ε, οδικέ μεταφορέ σε διεθνέ επίπεδο αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα λοιπόν σε συνεργασία και συμφωνία με τη γαλλική αντιπροσωπεία να υπενθυμίσω και να τονίσω κάποια σημεία για τα οποία θα αγωνιστούμε. Το πρώτο και κυριότερο, ε, αυτό στο οποίο θα επιμείνω περισσότερο, πρέπει στο πεδίο εφαρμογή των κρονισμων 1071 1071-2009 και 1072-2009 για τι συνθήκε πρόσβαση στην αγορά να συμπεριληφθούν και τα οχήματα που έχουν ε, μάζα μικρότερη των 3,5 τόνων, τα λεγόμενα ελαφρά φορτηγά. και πέραν των προσωπικών μου εμπειριών από την χρήση των οδικών δικτύων αλλά και με βάση μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο Φεβρουάριο. Αυτά τα, αυτά τα φορτηγά τα ελαφρά είναι το 80% των οδικών μεταφορών. Επομένως θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο και για λόγους ανταπροσωπευτικότητα αυτών των ε, ελαφρών φορτηγών να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού για να εξασφαλιστεί θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ όλων των ε, δραστηριοποιούμενων στο τομέα των μεταφορών. Επομένως πρέπει και αυτά τα φορτηγά να υπάγονται στις ίδιες συνθήκες με αυτές που ισχύουν για τα φορτηγά φορτίου άνω των 3,5 τόνων. Και επίσης ο 561 του 2006 ο οποίος αφορά τους χρόνους ανάπαυσης και εργασίας πρέπει να εφαρμόζεται και σε αυτά. Η ίδια μελέτη που σας ανέφερα νωρίτερα λέει ότι τα ελαφρά φορτηγά αλλά και τα δυο ταχύ αυτοκίνητα έχουν την ευθύνη για 94% των οδικών ατυχημάτων εναντί του 6% και 55% των, 58% ε, των οδικών ατυχημάτων οφείλονται σε κόπωση. Επομένως, είναι δυνατόν να λέμε ότι τα ελαφρά αυτά φορτηγά δεν τηρούν τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, δεν εφαρμόζουν τους κανόνες και μπορούν να αποτελέσουν μέσον στρέβλωσης του ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερα φορτηγά, αλλά και ταυτόχρονα αποτελούν τον τρόπο να εισαχθούν ή να να παραβιαστούν οι κανόνες για την ανάπαυση και την εργασία των οδηγών. Και με τον κύριο Μπαχ ε, έχουμε συζητήσει για την συμπερίληψη αντίστοιχα αυτών των ε, μικρότερων φορτηγών στην ε, οδηγία για τους χρόνους εργασίας και ανάπαυσης. Πρέπει επίση να περιοριστεί και σε αυτό συμφωνεί η Γαλλική Αντιπροσωπεία το περιθώριο τη διαμετακόμιση. Αυτό πρέπει να σημαίνει δηλαδή μία μόνο ένα μονοδρομολόγιο διαμετακόμισης κάθε τέσσερις μέρες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος του συστηματικού καμποτάζ. Να μην είναι νομάδες πλέον οι οδηγοί, να έχουν συνθήκες εργασίας αξιοπρεπείς, αντάξιε και τις αμοιβή του και τις υπηρεσίες που προσφέρουν και βέβαια με διαφύλαξη τη αρχή ελεύθερης κυκλοφορίας και ω εκπρόσωπο τη Γαλλική αντιπροσωπεία. θέλω να υπογραμμίσω ότι η αρχή της απόσπασης θα πρέπει να ισχύσει από την πρώτη μέρα της ε, διεθνού μεταφοράς εμπορευμάτων και στους οδηγούς ε, η οδηγία για την απόσπαση. Ο ταχογράφος μέχρι το 2023 μπορεί να είναι ευφυής ταχογράφος, μπορεί να διευκολύνει έτσι τους ελέγχους. Ψηφιακά λοιπόν δεδομένα πρέπει για μας να είναι απαραίτητα, πρέπει να είναι ο κανόνας για να εξασφαλίζουν και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωση στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη πρέπει να στηρίζονται στα υφιστάμενα εργαλεία ή τα όποια εμφανιστούν στη συνέχεια όπως ε, στην οδηγία για τη μη δηλωμένη εργασία και είμαστε υπέρ της ε, ε, γενικευμένης εξασφάλισης ελέγχων της ε, κατάργησης, της απαγόρευσης ουσιαστικά όμως των επιχειρήσεων που είναι μόνο γραμματοκιβώτια και ε, της εισαγωγή νομοθεσίας που δεν θα διευκολύνει την ύπαρξη και λειτουργία τους. Εκ μέρους λοιπόν της Γαλλικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα είμαστε κατά της, ε, του ανταγωνισμού και υποστηρίζουμε ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας. Ε, η ελεύθερη κυκλοφορία στην ενία αγορά δεν μπορεί να αποτελέσει πρόσχημα για να ε, καταρριφθεί καθέστηση εμπιστοσύνη, αμοιβέ εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών ή να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του πολίτη. Πρέπει ο εργαζόμενο στην Ευρώπη στι οδικέ μεταφορέ να τεθει σε κινδυνο η ασφαλεια του πολιτη πρεπει ο εργαζομενος στην ευρωπη στις οδικες μεταφορες να έχει αξιοπρεπεί συνθήκε εργασία Συνθήκε ασφάλειας τη χρήση του δρόμου. Τόσο ο ίδιος όσο και οι λοιποί χρήστε του οδικού δικτύου και βέβαια δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το ιδιαίτερα έντονο, τον ιδιαίτερα έντονο κινητικό χαρακτήρα, δηλαδή τη μεγάλη κινητικότητα των ε, οδηγών αυτών. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη γνωμοδότηση. Ε, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε μια φάση όπου μπορούμε πλέον να κρίνουμε τις ε, τροπολογίες. Βέβαια ο στόχος μας ε, είναι ακριβώς ο ίδιος, το να έχουμε αξιοπρεπείς ε, θέσεις εργασίας ε, και θέσεις απασχόλησης για τους εργαζόμενους και να έχουμε και σωστή αποζημίωση των εργανομένων. Υπάρχουν βέβαια κάποια θέματα όπου εγώ είμαι αναγκασμένος να τραβήξω μια κόκκινη γραμμή. Αναφέρομαι στην περίπτωση όπου συγκρούονται τα συμφέροντα των εργοδοτών με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Κάπως πρέπει εκεί να βρεθεί μια λύση. Ε, δεν ε, ζηλεύω την ε, εισηγήτρια, είναι πολύ δύσκολο το έργο της. Έχω πέντε ερωτήσεις να κάνω. Νομίζω ότι ανταγωνιστικότητα και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών δεν πρέπει να περιστούν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και αυτά τα λέω βεβαίως έχοντας κατά νου το θέμα της ε, κοινή αγοράς. Εξάλλου, εκείνο που πρέπει να επιδιώξουμε είναι να μειώσουμε το διοικητικό άχθος. η Ουγγρική αντιπροσωπεία τον ε, οδηγό δεν τον αντιμετωπίζει ως έναν αποσπασμένο εργαζόμενο, αλλά ως ένα εργαζόμενο που εργάζεται σε ένα κράτος μέλος. Βεβαίως, ε, παράνομες δραστηριότητες δεν πρέπει να συγχέονται με αθέμητο ανταγωνισμό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην κοινή αγορά να επιδιώξουμε καλύτερες συνθήκες ανταγωνισμού. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διεξάγουμε τον αγώνα κατά των ε, άδειλων εργαζομένων. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και θα μπορέσουμε να συμφιλειώσουμε τα διαφορετικά συμφέροντα. Επιτρέψτε μου να επισημάνω και κάτι άλλο, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε επ' αυτού. Δηλαδή, οι κανόνες, οι νομικοί κανόνες ε, τους οποίους εξετάζουμε νομίζω ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν όταν εφαρμοστούν για να μην υπάρχει χαός επόμενος ομιλητής. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρέικνα, τη σκιώδη για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Ε, νομίζω ότι ε, θα πρέπει από όλη αυτή τη συζήτηση να αφαιρέσουμε την συναισθηματική φόρτιση γιατί σε τελική ανάλυση δεν πρόκειται για να το λυδίσει, δεν είναι η σύγκρουση αυτή, αλλά πρόκειται για τις ελάχιστες απαιτήσει και στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους ανεξάρτητα από πού προέρχονται. Γι' αυτό λοιπόν εγώ στις ε, δικές μου τις ε, ε, τροπολογίες κατέστησα σαφή την προθεσή μου και εδώ στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Μεταφορών. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο όπου οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να επιβιώσουν και μακροπρόθεσμα μάλιστα στην κοινή αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χότσοβα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ξεκινώντας, ε, θέλω να πω ότι κατά την άποψή μου οι κανόνες πρέπει να είναι περισσότερο διαφανείς. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι οι διεθνείς μεταφορές και το διαμετακομιστικό εμπόριο δεν πρέπει να υπόκεινται στους ε, κανόνες περί απόσπασης εργαζομένων. Εάν βέβαια δεν συμφωνεί η πλειοψηφία, τότε ίσως θα πρέπει να είναι μικρότερο το χρονικό διάστημα από αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί το αντίθετο θα σήμαινε ότι περικόπτεται ε, το δικαίωμα της ελεύθερης παροχής μερσιών. Οι δύο ημέρες είναι υπερβολικές κατά την άποψή μου. Πρέπει να κάνουμε τους ε, σχετικούς υπολογισμούς. Εγώ έχω καταθέσει κάποιες ε, τροπολογίες και στηρίζω τις τροπολογίες ε, που προβλέπουν μία επιμήκυνση. Οι εννέα ημέρες ε, ε, που προτείνεται είναι ε, ικανοποιητικές, ίσως να είναι βέβαια λίγο υπερβολικές, αλλά κατά τα άλλα θα πρέπει να κάνουμε έναν σαφή υπολογισμό. Πρέπει να έχουμε κατά νου και το διοικητικό φορτίο των εταιριών μεταφορών. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τον υπολογισμό ηλεκτρονικά, επιγραμμικά. Έτσι λοιπόν να μπορεί ε, να γίνει υπολογισμό σε κάθε κράτος μέλος. Ο υπολογισμός αυτός ε, θα πρέπει να είναι προσπελάσιμος για όλους και μάλιστα δωρεάν. Μπας περιπτώσει, εγώ ε, θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, σαφήνεια των κανονισμών, ε, το διοικητικό βάρος θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερο γίνεται. Για μένα αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Ο κύριος Μπαχ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ, εγώ. να εκφράσω θερμές ευχαριστίες για το θέμα αυτό και την ε, περίπλοκο προς την εισηγητρία. Έχει προσπαθήσει να συνδυάσει όλες τις ιδέες. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Έχουν περιγράψει όλες τις δυσκολίες και ο Ζεγόμ εξήγησε πόσο αλληλένδετα είναι όλα. Μακρύ χρόνη οδήγηση, του οδηγού και ούτω καθεξής. Δύο είναι τα σημαντικά για μένα θέματα. Πρώτον, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να, απο, να αποκοπούν από την οδηγία για την απόσπαση οδηγή. Πρώτον και δεύτερον, πρέπει ξεκάθαρα να προσδιοριστούν οι κανόνες χωρίς να είναι περίπλοκοι οι υπολογισμοί. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Και γι' αυτό το επεσήμανε άλλωστε και η η συγγήτρια, το θέμα του καμποτάζ, της ε, διέλευσης, αλλά και στις διεθνείς μεταφορές νομίζω ότι πρέπει να ε, ζητήσουμε να είναι απλά τα μοντέλα. Είναι πολύ περίπλοκα αυτά τα οποία επιβάλλονται ως κανόνες στις ε, επιχειρήσεις. Πρέπει να είναι πολύ απλά και να ισχύουν από την πρώτη μέρα. Καλώς λίγο πρόεδρο. Ζώσες, είναι ο τελευταίος ομιλητής αυτό το γύρο και θα δώσω το λόγο στην κυρία Τλαμπάιωβα. Έχετε αρκετά, αρκετή δουλίτσα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως ακούσατε, είναι τόσο πολλές οι απόψεις, τόσο διαφορετικές εγώ θα ήθελα απλώ να ευχαριστήσω του σκιώδει συζητητέ και του υπόλοιπου συναδέλφου ε, για τη συνεισφορά του. Νομίζω ότι έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μα. Νομίζω όμω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Υπάρχουν ε, πολλά ε, σημεία ε, κοινά, όπως για παράδειγμα η έλεγχη, η επιβολή της νομοθεσίας και εκτιμώ ιδιαίτερος το γεγονός ότι όλοι κινείστε σε ένα πολύ επικοδομητικό πνεύμα και θέλετε να καταλήξουμε σε μια ρεαλιστική λύση όλοι μαζί. Και για να είμαι ειλικρινής, ελπίζω ότι μπορούμε να βρούμε μία λύση που να πηγαίνει πέρα από τον υπολογισμό ημερών, γιατί αν απλώς μιλάμε για έναν αριθμό ημερών, χάνουμε την ευρύτερη εικόνα ε, του προβλήματος. Και κάποιος μάλιστα εξημών ανέφερε από τη μία πλευρά την προστασία των εργαζομένων και από την άλλη την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Ε, κοιτάξτε, και εγώ θέλω να βρω μια ισορροπία μεταξύ των δύο. Δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα το ένα ή το άλλο. Πραγματικά θέλω να υπάρχει μια ισορροπία γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Οπότε όλοι οι συνάδελφοι που είπαν μόνο για την προστασία των οδηγών να σκέφτεστε και την ελεύθερη ε, ε, παροχή υπηρεσιών. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απολύτως με τα μέτρα επιβολής που πρέπει να είναι απλοποιημένα και συγκεκριμένα. Το υποστηρίζω αυτό γιατί πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει, μια, να υπάρχει κατάσταση αυθαίρετου ελέγχου και θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες ε, λεπτομέρειες για την περίπτωση του Τσέχου οδηγού ε, πάνω από χίλιους ε, οδηγούς στην Τσεχία που έχουν σκοπό να κάνουν αγωγή στους Γερμανούς ναι, αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι μόνο ένα ζήτημα κατώτατου μισθού. Είναι ζήτημα επιδομάτων επίση και ε, διαφορετικών συστημάτων και τη εναρμόνιση του πώ πληρώνεται ο καθένα σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Θέλει να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα. Και η εταιρεία μεταφορών που απασχολούσε τον Τσέχο οδηγό ήταν αυστριακή και κάθε προσπάθησε να ε, κάνει μήνυση στην αυστριακή εταιρεία και τελικά αυτή τον απέλησε. Οπότε στη συνέχεια ήρθε σε επαφή με τα συνδικάτα για να μπορέσει να κάνει αγωγή στη γερμανική εταιρεία. Τέλο πάντων, θέλω να πω ότι όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν, πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, γιατί μερικέ φορέ ε, αυτά τα μέτρα επιβολή ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες χώρες. Και θα ήθελα να πω ότι θα συναντηθούμε ήδη αυτή την εβδομάδα με τους σκιώδους συζητητές την Πέμπτη για να συζητήσουμε περισσότερο και ελπίζω να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο παρά το γεγονός ότι ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με την ψηφοφορία στη μήνυ Ολομέλεια αλλά ελπίζω και όλο το προσωπικό ε, να, ε, να είναι παρόν ε, να σας δώσω και μερικές επιλογές που έχω υπόψη μου και πριν από τη συνεδρίαση στους σκιώδους συζητητές εννοώ που προκύπτουν από τις τροπολογίες και από τις τοποθετήσεις των ομάδων, μας, των, ομάδων σας, των ομάδων σας. Ξέρετε, με ξέρετε πολύ καλά, ξέρετε πάρα πολύ πόσο επικοδομητική και ρεαλιστική θέλω να είμαι, οπότε σας παρακαλώ βοηθήστε με. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ψηφίσουμε στις 27-28 ε, Μαρτίου, στην Τραν 24 Μαΐου και δεν ξέρουμε ακόμη σε ποια ολομέλεια θα γίνει η ψηφοφορία. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα που αφορά βέβαια και πάλι αυτό το ζήτημα των μεταφορών και της κινητικότητας. Αφορά την τροποποίηση του κανονισμού 561-206 για τις ελάχιστες απαιτήσει ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο νέο χώρο οδήγηση, τα κατώτατα όρια για τα διαλύματα και τι περιόδου ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση και του κανονισμού 165 του 2014 για τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων. Δίνω το λόγο τώρα στον Ζωζ Μπακ. Θα ήθελα αυτή εξ αρχή να ευχαριστήσω του ε, συναδέλφου που έχουν καταθέσει τροπολογίες και οι οποίοι τάσσονται υπέρ τη ε, βελτίωση του τομέα μεταφορών, κυρίω υπέρ τη βελτίωση των συνθηκών εργασία των εργαζομένων, αλλά κυρίω επίση και για την οδική ασφάλεια. Όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ του. Χαίρομαι πάρα πολύ ε, είχαμε ήδη δύο συναντήσεις των σκιωδών και χαίρομαι που οι συνάδελφοι συμφωνούν μαζί μου ότι το βασικό πρόβλημα στην εφαρμογή των κανόνων ε, είναι ότι δεν υπάρχει συνεργασία. Είναι δύο δηλαδή βασικά τα προβλήματα. Και χαίρομαι που τώρα πλέον οι περισσότεροι επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι οι υπάρχοντες κανόνες ε, την χάνουν αναγνώρισης από τις επιχειρήσεις, από τους οδηγούς, από τις εποπτικές αρχές. Τέλος πάντων όλοι γνωρίζουν τώρα τους κανόνες, έχουν προσαρμοστεί και εγώ τα τελευταία χρόνια δεν έχω ακούσει συχνά να ε, λένε ότι κάποιοι επιτιμούν νέους κανόνες για το χρόνο οδήγησης. Εγώ ως εισηγητής ε, πρόκειται να επεξεργαστώ την ε, εισήγησή μου και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα τη στηρίξουν βέβαια όλοι, Υπότιτλοι πολύ και θέλω να πιστεύω ότι και θα εισακουστεί η άποψή μα ε, στην Επιτροπή Μεταφορών γιατί αυτό είναι το επόμενο καθήκον μα. να παρουσιάσουμε τη γνωμοδότησή μα στην Επιτροπή των Μεταφορών. Θέλω να θίξω και κάποια θέματα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έθιξαν αρκετοί συνάδελφοι. χρόνο αναφορά ε, τεσσάρων εβδομάδων όπου οι οδηγοί μπορούν να εργάζονται 180 ώρε και να τι ε, κατανέμουν στις τέσσερις εβδομάδε. Κόκκινη γραμμή για μένα, απαράδεκτο. Αυτό θα επιδεινώσει τη θέση των οδηγών και θα ε, θέσει και σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Τα τελευταία χρόνια ο συνάλφος Ζερόμ Λαβριέ επισήμανε ότι έχει ε, προκύψει ένα άλλο επιχειρηματικό μοντέλο και υπάρχουν νέα μικρά επαγγελματικά οχήματα. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ αριθμητικά. Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτά πρέπει απαραίτητα να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Από ποιο βάρος, σε ποια ακτίνα ή αν θα, έχουν, αν θα είναι εξοπλισμένα με ταχογράφους ή όχι, πότε θα γίνουν αυτά, πώς θα γίνουν αυτά, αυτά βέβαια τα συζητάμε αυτή τη στιγμή. Το περίφημο, η περίφημη απαγόρευση να κοιμούνται οι οδηγοί στην ε, καμπίνα. Αυτό δεν ξέρω αν είναι σωστό, γιατί δεν υπάρχουν αρκετές ε, θέσεις και χώροι στάθμευσης, ούτε και ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να ορίσουμε μια καταληκτική ημερομηνία και να δουλέψουμε σωστά. Είμαι συγητή και για την Ευρωβινιέτα. Εκεί λοιπόν ε, θα, προσθε... θα προσπαθήσω τα έσοδα που θα προκύψουν για τις υποδομές αυτά να επενδυθούν ε, σε θέσεις ε, απασχόλησης ε, και ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής. Περίπλοκο το θέμα. Υπάρχει και το θέμα του χρόνου ανάπευσης των οδηγών που επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Νομίζω ότι από αυτού έχουμε ήδη συζητήσει. Πρέπει να ερμηνεύσουμε, να ορίσουμε τι σημαίνει ιδιωτικός χώρος. Πρέπει οι ορισμοί να είναι απολύτως απολύτως σαφής, γιατί επαναλαμβάνω η βασικότερη κριτική που ασκείται στον ισχύοντο κανονισμό είναι η ασάφεια. Επιτρέψτε μου και δύο τελευταία θέματα. Ο βασικός μας στόχος ε, είναι ε, να σταματήσουμε, να δώσουμε τέλος σε αυτό το νομαδικό τρόπο ζωής των οδηγών. Και νομίζω ότι ε, και οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τα χρονοδιαγράμματα, καταρτικά αρκετά έγκαιρα. Πρέπει λοιπόν να είναι δυνατόν οι ε, χρόνοι οδήγησης ε, να έχουν μορφωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο οδηγός να μπορεί να επιστρέψει στην κανονική του κατοικία χωρίς ε, αυτό το γεγονός να επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα της επιχείρησης. Κατά τα άλλα πρέπει και να βελτιωθεί το κύρος του οδηγού, να είναι πιο ελκυστικό το επάγγελμα αυτό για να μην υπάρχει έλλειψη εργαζομένων Κάτι τελευταίο για τους ευφυείς ταχογράφους. Όσον αφορά το θέμα αυτό, οι προβλεπόμενες προθεσμίες είναι απαράδεκτες για μένα. Τα 15 χρόνια είναι γελία θα τα χαρακτήριζα. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να περιορίσουμε αυτό το χρονικό διάστημα, γνωρίζοντας βέβαια ότι η εγκατάσταση και η αναδρομική, ο αναδρομικός υπολογισμός προκαλούν σημαντικές δαπάνες. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρχει ε, μια λογική μεταβατική περίοδος. Γίνεται λόγος για το 21 μέχρι το 23. Πέρα από το 23, το 34 ας πούμε, αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους και χαίρομαι για την συνέχιση αυτής της συνεργασίας. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Κρίστενσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πάρα πολύ καλή συνεργασία ε, και τους κοιόδης εισηγητές. Ε, έχουμε την ευθύνη να βρούμε λύσεις ε, που δημιουργούν γέφυρες μεταξύ των πολύ διαφορετικών θέσεων. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η βασική προτεραιότητά μου, οι βασικές προτεραιότητές μου είναι οι εξή. Η, περίοδο αναφορά, η περίοδος αναφοράς θα έπρεπε να παραμείνει στις δύο εβδομάδες όπως ισχύει αυτή τη στιγμή. Η επέκταση ανάπτυξή τη θα είχε αρνητικό αντίκτυπο και για τις κοινωνικές συνθήκες αλλά και για την οδική ασφάλεια. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι οδηγοί δεν περνάνε τον εβδομαδιαίο του χρόνου ανάπαυση στην καμπίνα αλλά στο σπίτι τους ή σε αξιοπρεπή καταλήμματα τα οποία θα παρέχει ο εργοδότης. Η χρήση η πρακτική της νομαδικής ζωής πρέπει να σταματήσει, πρέπει να έχουν μια εγγυημένη δυνατότητα να επιστρέψουν στις οικογένειές τους τουλάχιστον κάθε τρίτη εβδομάδα. Ε, επίσης ε, πρέπει να σέβονται τους ε, κανόνες όταν κάνουν οδικές μεταφορές διεθνείς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παραθυράκι στην ομοθεσία και αυτό πρέπει να το καλύψουμε. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, πρέπει να υπάρξει πλήρης εφαρμογή των εφιών ταχογράφων το συντομότερο δυνατόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πραγματική εφαρμογή των κανόνων που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να θεσμοθετήσουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε μια ε, επικοδομητική συνεργασία. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ΣΥΑΡ είναι κανείς εδώ? Όχι. Για τους φιλελεύθερους η κυρία Τλαμπάγιοβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ και, στους τρεις, ε, και στα τρία θέματα είμαι, είμαι, ασχολούμαι και με τα τρία θέματα, είμαι σκιώδης συγγήτρια και τα άλλα δύο. Πραγματικά θαυμάζω πάρα πολύ τους ε, εισηγητές γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυάσει κανείς και ε, τα τρία αυτά θέματα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μπακ για την οργάνωση των σκιο... συνάντηση των σκιωδών εισηγητών την περασμένη εβδομάδα. Ε, ελπίζω ότι θα έχουμε άλλη μία κατά τις ερχόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το, πρώτο... για το σχέδιο συμβιβαστικών τροπολογιών. Πολλά πρέπει να συζητήσουμε, πολλά επίμαχα ζητήματα. Να αναφερθώ σε μερικά. Νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, ε, στους συμβιβασμούς ε, το ότι πρέπει να είναι θετικός ο αντίκτυπος των κανόνων ότι θα βελτιώσουν τις ε, συνθήκες εργασίας των οδηγών αλλά παράλληλα δεν δυσχεραίνουν εντελώς το έργο των επιχειρήσεων. Για την ώρα βασική μου ανησυχία είναι η εβδομηδιαία ανάπαυση των οδηγών, συμβαστική τροπολογία 15. Υπάρχει έλλειψη ασφαλών θέσεων στάθμευσης και έλλειψη ασφαλών καταλημάτων στου αυτοκινητοδρόμους στην Ευρώπη και πολύ αμφιβάλλω κατά πόσο μπορούμε στην πράξη μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτόν τον περιοριστικό κανόνα ακόμη και αν φαίνεται ένα ηρωικό βήμα ε, για να επιτρέπεται στους οδηγούς ε, να έχουν μια ιδιωτική, ένα ιδιωτικό κατάλημα που θα είναι φιλικό προς το ε, φίλο τους, έτσι λέει τουλάχιστον συμβαστική τροπολογία. Δύσκολο μου φαίνεται αυτό. Ε, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στις ανησυχίε των εισηγητών ε, για, την, ε, για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα κάτω των 3,5 τόνων. Καλό θα ήταν να έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία, κάποια δεδομένα, κάποια αποδεικτικά στοιχεία που να ε, που να δικαιολογεί τη συμπερίληψη των ε, οχημάτων αυτών ε, στον 561 του 2016. Το έχουμε ξαναπεί στη συνάντηση των σκιωδών και θα το ξαναπούμε. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τους οδηγούς και τις εταιρείε για το διακανονισμό του χρόνου εργασίας τους, όχι βέβαια ώστε να, μειωθούν, να μειωθεί η ποιότητα των συνθήκων εργασίας των οδηγών, αλλά μπορούν να αρχίζουν ε, από τις περιφερειακές περιοχές ε, ε, το ταξίδι τους. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, ε, μπορεί να υπάρχουν μποτιλιαρίσματα, μπορεί να μην υπάρχουν ε, τα κατάλληλα καταλήματα για να ξεκουραστούν. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε μια σχετική ευελιξία, να δούμε υπό ποιε συνθήκες και πότε πρέπει να γυρνά πίσω στην, στο σπίτι του ή σε κάποιο μέρος επιλογής του οδηγός. Κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι πρέπει να αποζημιώνονται αυτά τα ταξίδια από, τους, από τις επιχειρήσεις. Όμως ε, αυτό ρυθμίζεται από την οδηγία απόσπασης ε, εργαζομένων και θα ήταν καλό να μην αναφέρουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση τέτοιου είδους ε, ρυθμίσεις. Με χαρά όμως αναμένω την επικοδομητική συνεργασία μας κατά τις ερχόμενες ημέρες και σε εβδομάδες και θα προσπαθήσω όπως και για τη δική μου έκθεση να είμαι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική και επικοδομητική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόπες Βερμέιο, Γκουε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του και την προσπάθεια πάνω απ' όλα να εξασφαλιστούν συμβαστικές λύσεις για τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας των εργαζομένων. είναι πολύ σημαντικό να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες ε, στην οδική ασφάλεια αυτών των ε, συνθήκων εργασίας. Είναι σωστός ο δρόμος που έχουμε ακολουθήσει. Το συμφέρον του εργαζομένου πρέπει να είναι κύριος ε, γνώμονας μας. Αυτοί είναι που εργάζονται, που οδηγούν. Πρέπει να γυρίσουν σπίτι τους ασφαλείς όταν θα έχουν διασχίσει τους δρόμους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν πρέπει να δοθεί έμφαση. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι συμφωνούμε ως προς την τήρηση των ε, εβδομαδιαίων ορίων για την οδήγηση και των ελάχιστων ορίων στάσης και ανάπαυσης. Όπως επίσης και, κάλυψη, και την κάλυψη των εξόδων επαναπατρισμού του οδηγού από την επιχείρηση. Αλλά αυτά δεν αρκούν. Οι κανόνες δεν αρκούν γιατί πρέπει να εφαρμοστούν κιόλας. Είναι σημαντικό λοιπόν να ενσωματωθεί το ταχύτερο δυνατό στα φορτηγά ο ευφυής ταχογράφος, πάντως όχι πιο αργά από το 2021. Πρέπει να είναι εγκαταστημένο σε όλα τα φορτηγά, να είναι ευχερής ο έλεγχος. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. που με ενδιαφέρει για να τονίσω και τις θέσεις μας πρέπει να αποφύγουμε τις παρεκκλήσεις όταν μιλούμε για ελαφρέα φορτηγά. Αυτά μπορούν να αποτελέσουν ε, ένα κίνδυνο για παραθυράκια ή κενά στον νόμο αν δεν καλυφθούν. Όπως επίσης ε, εάν δεν καλυφθούν οι οδηγοί των μη επαγγελματικών φορτηγών, δηλαδή οδηγοί που οδηγούν το ιδιόκτητο φορτηγό ανεξαρτήτως ε, φορτίου πρέπει και αυτοί να καλύπτονται γιατί παραμένουν οδηγοί. Πρέπει αυτό να καλυφθεί λοιπόν, να συμπληρωθεί στο κείμενο. Θα μας απασχολήσει βέβαια σε επόμενες ημέρες, θα το επεξεργαστούμε και επαναλαμβάνω τη βούλησή μου για συνεργασία σε συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντέλη για τους πράσινους. Πρόεδρε ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Ζόρζ, Καταρχάς θέλω να σας ε, συγχαρώ ως εισηγητή για την εξαίρετη αυτή έκθεση, πληρέστατη. Και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι πράσινοι έχουν καταθέσει ελάχιστες τροπολογίες στην έκθεσή σας. Όπως και εσείς, είμαι και εγώ κατά της επέκτασης της περίοδου αναφοράς που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που θα έχει, το έχω επισημάνει και το ξαναλέω, αρνητικά, ε, αρνητικές συνέπειες στο χρόνο εργασίας και στο λέω ως Πρόεδρος της Επιτροπής των Μεταφορών. Το θέμα της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές κρίνεται από αυτό. Επίσης, συμφωνώ μαζί σας και βέβαια με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου περί απαγόρευσης της εβδομαδιαίας ανάπαυσης στο φορτηγό μέσα, στην καμπίνα του φορτηγού η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ αντιβαίνει, το λέω ξεκάθαρα, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, διότι εάν αύριο αν επιτραπεί αυτό, οποιαδήποτε άλλη λύση προταθεί αύριο θα είναι εκτεθειμένη σε αφισβήτηση και προσφυγέ. Και βεβαίως είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε την ε, απόλυτα σαφή νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Χαίρομαι που οι τροπολογίες μου σχετικέ με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασίας έχουν συμπεριληφθεί ήδη στην πρώτη έκδοση των συμβαστικών τροπολογιών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν επιλεκτική εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μπορούν με τους ελέγχους να αντιμετωπιστούν. Το ευρωπαϊκό δηλητήριο που κάνει κακό στο ευρωπαϊκό όραμα είναι το κοινωνικό dumping. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε πλέον να πάψουμε να είμαστε υποχρεωμένοι κάθε χρόνο να συζητούμε το τι θα κάνουμε αν δεν ισχύουν οι έλεγχοι και αν δεν γίνονται οι έλεγχοι όπως πρέπει. Πρέπει αυτή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, γιατί είναι πραγματικά μοχλός κινητήριος για το έργο αυτό να ε, επιληφθεί, να θεσπιστεί και να επιληφθεί αυτού του θέματος για τις οδικές μεταφορές. Και αυτό θα αποτελέσει τεράστια πρόοδο και πολύ πολύ σημαντικό μήνυμα ένα μήνυμα το οποίο ζητούν και απαιτούν και όλοι οι μεταφορείς αλλά και όλα τα κράτη-μέλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σα καλέσω τι τροπολογίε αυτέ να τις εξετάσετε με μεγάλη προσοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει ψήφισμα μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, σύσταση της ε, υπηρεσίας αυτής το Μάρτιο. Με την ευκαιρία αυτή είναι απαραίτητο να δηλώσουμε απερίφραστα ότι την ε, υπηρεσία αυτή την υποστηρίζουμε και η Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή των Μεταφορών. Ένα άλλο κεντρική σημασία θέμα, πολύ σημαντικό επίσης, είναι η επιτυχία στην υλοποίηση της οδηγίας. Έχουμε το θέμα του εφιούς ταχυκογράφου και βεβαίως μπορεί κανείς να συζητήσει πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και μέχρι πότε να έχει εισαχθεί ο ταχογράφος. Εγώ θα πω 2022. Όπως και να έχει όμως θα είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από το 2034. Γιατί το κοινωνικό ντάμπινγκ ε, θα έχει περιθώριο να πολλαπλασιαστεί. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι λοιπόν. Πρέπει να αποστείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα για, με τις εκθέσεις αυτής προς τα έξω και να αποδείξουμε ότι δεν θέλουμε να φέρουμε αντιμέτωπους ε, εργαζομένους του ενός κράτους ε, με εργαζομένους του άλλου κράτους, αλλά ότι μέλημά μας είναι η υγεία και η ασφάλεια όλων των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές από όλες και σε όλες τις χώρες τη Ευρωπαϊκή Ευρω... Ευρωπαϊκής Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητάει κανεί από του EFDD. Ο κύριο Μαχτάν, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Μόνο 13 τροπολογίες έχουμε καταθέσει και αυτό δείχνει πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από τη δουλειά σας και μάλιστα ευχαριστούμε για το εικόνσο ότι η πρόταση και το ανέφερε και ο κύριος Λαβρίγιο νωρίτερα πολύ σωστά για τα ελαφρά φορτηγά που έχουμε κάνει και εμείς έχει γίνει δεκτή πρόκειται για μια σαφή στρέβλωση της νομοθεσίας είναι σαφώς καλύτερο το όρο των 200 από αυτό των 100 χιλιόμετρων επίσης ευχαριστούμε για την ενσωμάτωση της υποβάθμισης των κανόνων για την ανάπαυση στους τέσσερις εβδομάδες σε σχέση με αυτό ε, που πρότεινε η Επιτροπή που ήταν υποβάθμιση Επίσης ένας οδηγός θα πρέπει να μπορεί να επιστρέφει στο σπίτι του μία φορά τη βδομάδα τουλάχιστον για να αναπαύεται και όχι μια φορά το μήνα όπως ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε περιορισμό στην ανάπαυση θα πρέπει να ίσως και λύσετε μέχρι το τέλος της ακόλουθης εβδομάδας. Και είμαι πολύ σύντομο γιατί κάνατε εξαιρετική δουλειά στην αρχή αυτής της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, και εγώ ε, θεωρώ ότι αυτά τα τρία έγγραφα θα πρέπει να εξεταστούν ε, από κοινού. Και δεν θα ήθελα βέβαια να επαναλάβω αυτά τα οποία είπα για το πρώτο έγγραφο, όσον αφορά στο κοινωνικό dumping και επ' αυτού ισχύει η άποψή μου, αυτά που είπα προηγουμένως. Νομίζω και άλλοι συνάδελφοι επισήμαναν το κοινωνικό dumping. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι όλα αυτά δεν θα πρέπει να τα μπερδεύουμε με παράνομους και λαθρεεργαζόμενους ε, απασχολούμενους το κείμενο μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε το θέμα της, ε, του εβδομαδιαίου χρόνου ανάπαυσης, αλλά το όλο το σύστημα ε, θα είναι ευέλικτο μόνο εάν πέρα από το χρόνο διήγηση, επανεξετάσουμε και το χρόνο της ανάπαυσης. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θέματα ε, πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. 45 ε, ώρες την εβδομάδα ως χρόνο ανάπαυσης. Ε, αυτές οι 45 ώρες δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι τους ε, ευρωπαϊκούς δρόμους δεν υπάρχουν φυλασσόμενοι χώροι στάθμευσης και ικανοποιητικά καταλήματα. Πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες, ε, παραδείγματο χάρη, του να κάνει κανείς ε, ένα μπάνιο. Έχω μιλήσει με μεταφορείς και μου είπαν ότι στη Γερμανία Υπάρχουν μόνο 352 ε, χώροι στάθμευση και σε αυτούς μόνο οι 13 χώροι είναι φυλασσόμενοι και προσφέρουν τη δυνατότητα καταλήμματος, τη δυνατότητα μπάνιου και όλα τα απαραίτητα. Μόνο 13. Εγώ λοιπόν ε, θέλω να επισημάνω ότι στην ε, Ουγγαρία οι ασφαλιστικές εταιρείες ε, δεν θα είναι πρόθυμες να ασφαλίσουν αυτοκίνητα αν ο οδηγός ε, δεν βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουν αυτοκίνητα μόνο εφόσον αυτά παραμένουν και σταθμεύουν σε φυλασσόμενους χώρους στάθμευσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπαχ. Πάρα πολύ σύντομος θα είμαι. Ευχαριστώ πολύ τους ε, συναδέλφους ε, για τις παρατηρήσεις που έκαναν, για τις προτάσεις τους. Επιτρέψτε μου, ε, τονίσω και εγώ δύο-τρία πράγματα. Η συνάδελφος Μαρτίνα, πολύ σωστά νομίζω, επισήμανε τα στατιστικά δεδομένα, ε, το ότι λείπουν κάποια στοιχεία, ε, το πώς εξελίσσονται οι μεταφορές με τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Θέλω όμως να σας πω ότι αν αυτή τη στιγμή μιλάμε για 1, 2, 3% αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θεωρώ ότι το δικό μας το καθήκον ως υπεύθυνη πολιτική είναι να επιδείξουμε οξυδέρκεια, να προλάβουμε εξελίξεις. Δεν επιτρέπεται εκ των υστέρων να προσπαθούμε να μπαλώσουμε τα πράγματα και μόνο τότε να προσπαθούμε να νομοθετούμε. Υπάρχει αυτό το μοντέλο που εγώ το βρίσκω ιδιαίτερα προβληματικό ε, τόσο για τους απασχολούμενους όσο και για την οδική ασφάλεια. Ε, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα ε, μέχρι να φτάσουμε στον πλήρη εκφυλισμό. Και κάτι άλλο κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά στους χώρους στάθμευσης, νομίζω ότι όχι μόνο σε αυτήν την έκθεση, αλλά γενικότερα θα πρέπει να ε, εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, να ασκήσουμε πίεση για να υπάρχουν φυλασσόμενοι χώροι στάθμευσης. Ξέρω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να γίνει εν μια νυχτή, αλλά σε πολλά κράτη-μέλη οφείλουμε να επισημάνουμε το πρόβλημα. Για μένα πραγματικά είναι υπερβολικό το να ζητάει κανείς από τον οδηγό τη νύχτα που υποτίθεται ότι ξεκουράζεται να ελέγχει, να είναι και υπεύθυνο για το εμπόρευμα. Αυτό πραγματικά είναι ακραία υπερβολή. Δεν τι κάνουμε εμείς. Για φανταστείτε, όταν τελειώνουμε εδώ τη δουλειά μας, μετά να έπρεπε να είμαστε και φύλακες ε, οποιοδήποτε πράγματος. Αυτό το βρίσκω υπερβολικό ε, ως απέτηση και από τις ασφαλιστικές εταιρείε, αλλά και από τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα λοιπόν για το χρονοδιάγραμμα. Εδώ 27-28 Μαρτίου, 24 Μαΐου στην Τραν, και για την Ολομέλεια θα προσδοριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο και θα πρότεινα να συνεχίσουμε αυτή την ε, παράλληλη εξέταση και τη συνεργασία με την Επιτροπή των Μεταφορών. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η τροποποίηση του κανονισμού 1071-2009 και του 1072-2009 με σκοπό την προσαρμογή του στις εξελίξεις του τομέα. Η κυρία Λαπεφοντανιέ, η συγκεκριά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα, μια χρονομοδότηση η οποία παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες, 273 ε, τροπολογίες, πολλές αντιφατικές ε, απόψεις. Ε, έχω στείλει ένα πρώτο σχέδιο των τροπολογιών των συμβιβαστικών. Ήδη από σήμερα, αύριο το πρωί θα γίνει μια πρώτη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Έχουμε, ήδη έχουμε κάνει μια συνάντηση έτσι, διερευνητική. Είναι πολύ δύσκολο πάντως γιατί στην ουσία κάποιες τροπολογίες είναι εντελώς αντιφατικές όμως είμαι αισιόδοξη και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Είμαι πεπισμένη ότι θα καταφέρουμε να βρούμε έναν πραγματικό συμβιβασμό. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στις πτυχές που μου φαίνονται πλέον προβληματικές σε σχέση με τις τροπολογίες που έλαβα όσον αφορά τα ελαφρά οχήματα. Όπως το γνωρίζετε, πρόκειται για οχήματα κάτω των 3,5 τόνων και δεν καλύπτονται από τον 1071 κανονισμό. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ το θέμα των ε, ψευτοαπασχολουμένων και των εταιριών ε, γραμματοκιβωτίων ε, που υποτίθεται ότι απασχολούν αυτούς τους ψευδείς ελεύθερους επαγγελματίες. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω να δημιουργήσουμε τεράστια εμπόδια ώστε να δυσκολεύει η κατάσταση και των επιχειρήσεων στον τομέα. Πολλές τροπολογίες ισχυρίζονται ότι κάποιες διεθνείς μεταφορές πρέπει να εξαιρούνται. Συμφωνώ με την τροπολογία 32 του George Μπακ, δηλαδή ότι Υπάρχει μία εξαίρεση για τα οχήματα από 2 ως 3,5 τόνους και όσον αφορά τώρα τις ε, οικονομικέ απαιτήσει, νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες απαιτήσει ε, ε, με τα πολύ μεγάλα φορτηγά. Ε, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι γιατί διαφορετικά θα υπάρξει αρνητικό αντίκτυπος ε, στην εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερικής αγοράς αλλά και στην αγορά των μεταφορών. Όσον αφορά λοιπόν τις επιπλέον απαιτήσει των κρατών μελών ε, για την άσκηση των, του επαγγέλματο του οδηγού οι περισσότεροι ζητούν να διατηρήσουμε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του κανονισμού του 1071 που, να, που, λέει δηλαδή ότι πρέπει τα κράτη, οι μέλη πρέπει να θέτουν επιπλέον ε, περιορισμούς. Συμφωνώ. Η ελευθερία εγκατάστασης. Φυσικά αυτό είναι θεμέλιος λήθος της αγοράς, ε, της εσωτερικής αγοράς. Ε, είναι απαραίτητο λοιπόν από τη μία να εξασφαλίζουμε αυτή την ελευθερία και από την άλλη να σεβόμαστε τα κριτήρια που ισχύουν. Ώστε, θα, ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις αθέμητες πρακτικές που αυτή τη στιγμή συνιστούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Όσον αφορά τώρα τα κριτήρια που επιτρέπουν την αξιολόγηση ε, πιστεύουμε ότι η, οδηγία περί απόσπασης δεν μπορεί να θεωρηθεί κριτήριο γιατί πρόκειται για άλλους εργαζόμενους. Όμως μπορούμε να καταλάβουμε ότι όντως συμπεριλαμβάνουμε τους κανόνες που ε, έχουν να κάνουν με το καμποτάζ ε, γιατί Ο κίνδυνο είναι ένα ενδεχόμενο πρόβλημα για την ε, εσωτερική αγορά. Ναι, το Καποτάζου είναι πράγματι το πιο επίμαχο ζήτημα και είναι πολύ αντιφατικέ οι απόψει. Ε, το κεφάλαιο 3 του 1072 είναι πολύ σαφέ. Υπάρχουν τροπολογίες που ζητούν τη μείωση του αριθμού των ε, μεταφορών και άλλε που ζητούν την αύξηση. Λοιπόν, αυτό που νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι να μην επιστρέφουν κενά τα φορτηγά σιγά άδεια μετά από μια τέτοιου είδου μεταφορά. Ο αριθμό των ημερών πρέπει να είναι επαρκή, ώστε οι μεταφορεί να μπορούν να ε, διεκπεραιώνουν την αποστολή του και να μπορούν να γυρίσουν στο κράτος μέλο του και στο σπίτι τους που είναι επίση αυτό πολύ σημαντικό. Η επιστροφή της της, ε, στη χώρα, ε, στο κράτο μέλος εγκατάστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα των ελέγχων είναι επίσης σημαντικό όσον αφορά την επιβολή του κανόνα για τους αποσπασθέντες ε, όσον αφορά το καμποτάζ. Εγώ διαφωνώ και δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε αυτό το ζήτημα να το καλύψουμε με το lex specialis μόνο αυτό το ζήτημα. Για τα υπόλοιπα ευχαρίστω να μιλήσουμε, να διαπραγματευτούμε, να φτάσουμε σε ένα κείμενο το οποίο βέβαια θα είναι αντικείμενο υποστήριξη όλων των συναδέλφων. Αύριο το πρωί λοιπόν θα έχουμε την πρώτη συνάντηση σκιωδών ε, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ε, Σιμό. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σάιμον, συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνετε, συνάδελφοι, όλοι σας και όπως ε, υπόθηκε υπάρχει μια, ένα τεράστιο φάσμα απόψεων. Νομίζω για το καμποτάζ τουλάχιστον υπάρχουν 15 διαφορετικά μοντέλα που προτείνονται στις διάφορες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί ως τώρα οποίες δεν είναι μόνο 15 διαφορετικές τροπολογίες, αλλά καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα ε, θεώρησης του, του ζητήματος. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να πω πάρα πολλά σήμερα, γιατί πιστεύω ότι εν ώψη της ε, συνάντησης των σκιωδών αύριο δεν είναι πολλά αυτά που θα μπορούσα να πω σήμερα και που να είναι ε, πολύ πολύτιμα. Ο συνάδελφος είπε ήδη πολλά. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση γιατί υπάρχουν τόσο πολύ διαφορετικές απόψεις, αποκλίνουσες. Όλοι μιλούμε για το πόσο περίπλοκο είναι αυτό το ζήτημα. Ε, ας αρχίσουμε λοιπόν και τις διαπραγματεύσεις. Σύντομα όμως, θα ήθελα να σημειώσω, δεν έχουμε δει τις συμβιβαστικές τροπολογίες ακόμη, μόλις, μόλις τις λάβαμε αλλά δεν τις έχουμε ε, διαβάσει ακόμη όλα αυτά θα γίνουν μέχρι αύριο. Είναι όμως ε, χρήσιμο να σημειώνει κανείς ε, σε σχέση με τα τρία αυτά θέματα που εξετάζουμε από κοινού. Να μην ξεχνούμε ότι είναι ένα από τα τρία που δεν είναι μία αρμοδιότητα κοινή της δική μας Επιτροπής και της Επιτροπής Μεταφορών. Είναι δική μας γνωμοδότηση ε, προς την ΤΡΑΝ και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί για το τι μπορούμε να πετύχουμε εμείς ως Επιτροπή Απασχόληση Να γνωρίζουμε λοιπόν πολύ καλά ε, ποια είναι η θέση της αρμόδιας επιτροπής που είναι η Επιτροπή Μεταφορών για το Καποντάζ. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι με τις τροπολογίες μας διατηρούμε τον ε, τρέχοντα ορισμό για, τους, ε, για το καποντάζ και ότι υπάρχει ένας περιορισμός 48 ώρων ε, μετά την τελευταία μεταφορά αυτή είναι και η γραμμή του εισηγητή των σοσιαλδημοκρατών στην Επιτροπή Μεταφορών. Υπάρχει, όπως είπα, όμως τεράστιο φάσμα διαφορετικών απόψεων από τους συναδέλφους. Όσον αφορά την πρόσβαση τώρα, ε, είμαστε πολύ σαφείς, ε, τα ελαφρά οχήματα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα τέσσερα κριτήρια πρέπει να ισχύουν κατά τη γνώμη μας και στα ελαφρότερα οχήματα και είναι σαφές από τις τροπολογίες ότι πολλοί δεν θα ήθελαν να ισχύσει κάτι τέτοιο. Ε, για τη χώρα εγκατάστασης, εδώ υπάρχει κάποια μορφή συμφωνία. Δεν θα χρειαστεί ενδεχομένως να μιλήσουμε πολύ γι' αυτό αύριο. Νομίζω ότι διαφωνούμε ή τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει αν διαφωνούμε στο να προσθεθεί το καμποτάζ στον κανόνα των παραβάσεων, αλλά εμείς έχουμε υποβάλει τροπολογίες που να προτείνουν ένα κοινωνικό ε, ταμείο εγγύησης ε, στο κομμάτι που αφορά την πρόσβαση ε, από ό,τι γνωρίζω έχουν ε, υποβάλει συνάδελφοι για περιόδους ανάπαυσης διαφορετικές μετά από το καμποτάζ. Όλα αυτά ε, θα αρχίσουμε να τα συζητούμε σε περισσότερη λεπτομέρεια αύριο. Κάποιες ε, σύντομες ερωτήσεις λίγο περισσότερη σαφήνεια θα ήθελα ως προς το εξής. Είπατε εσείς ως εισηγήτρια μας ε, ότι, ότι υπάρχουν τροπολογίες που προτείνουν Το κομμάτι δηλαδή που έχει διαγραφεί από το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτό που αφορά τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα και μιλάει για την ε, ε, για τον τζίρο των τελευταίων ετών. Ε, των τελευταίων ετών. Εγώ δεν το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Δεν κατάλαβα αυτή την τροπολογία που ζητά αυτή τη διαγραφή. Κάποιο δεν θέλει, εντάξει, τη γραφειοκρατία που είναι άχρηστη. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρο ε, τι ακριβώς, ε, σε τι ακριβώ αφορά η γραφειοκρατία αυτό το ζήτημα. Αυτό το θέμα του Lex Specialis που το είχαμε συζητήσει και την, προηγούμενη φορά, άκουγα, αλλά ακόμη δεν, είμαι βέβαιος ότι έχω καταλάβει καλά τι, τι ακριβώς εννοείται. Η συγγήτρια μίλησε για την πρότασή σας. Μήπως μπορείτε κάποια από εσά να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις σε σχέση με τις συνέπειες της προσέγγισης αυτής για το θέμα μας, γιατί πραγματικά αγωνίζομαι να καταλάβω. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Στέβενς. ECR. Σας ευχαριστώ πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνώ απολύτως με την εισηγήτρια όσον αφορά την καταπολέμηση των εταιριών ε, γραμματοκιβωτίων Πρέπει να είναι η κύρια προτεραιότητά μας. Η παροχή βεβαίως υπηρεσιών είναι διαλύθος του συστήματος των μεταφορών, αλλά οι παράνομες δραστηριότητες την ε, οδηγούν, ε, την εκθέτουν σε σημαντικούς κινδύνους. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέψουμε να υπάρχουν τέτοιου είδου επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που συστήνονται σε κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν διαρκείς δραστηριότητες. Και γι' αυτό χρειάζεται μια ατομική αξιολόγηση πιστεύω ε, λαμβανομένων υπόψη διαφόρων ε, στοιχείων, καλύτερη έλεγχη, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να καλυφθούν τα κενά στο νόμο και η διαμετακόμιση θα πρέπει να ανταποκρίνεται και στους περιβαλλοντικούς κανόνες. Δεν μπορεί δηλαδή η διαμετακόμιση να αποτελέσει πρόσχημα για να απαλλαγεί κανείς από την τήρηση των κοινωνικών κανόνων στη χώρα υποδοχής. Δεν είμαι υπέρ του τύπου φιλελευθεροποίησης, ε, απελευθέρωση καλύτερα της αγοράς που προβάλλεται εδώ. Προτείνω τον περιορισμό σε τρεις μέρες προτείνω κανόνες ευχερείς στην εφαρμογή του και βεβαίω ε, προσβλέπω στη συνεργασία με την εισηγήτρια και του κοιόδης εισηγητέ για να καταλήξουμε σε ένα καλό και ισορροπημένο κείμενο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φιλελεύθερη, κυρία Τσιλαμπάτοβα. Ναι, <laughs> πάλι εγώ. Και ευχαριστώ πολύ Βερόνικα για την παρουσίαση. Περιμένω με ανυπομονησία την πρώτη μας συνεδρίαση σκιωδών που θα λάβει χώρα αύριο. Θα ήθελα να απαντήσω και στον κύριο Σάιμον, γιατί αν κατάλαβα καλά το ερώτημα και ίσως να αφαιρέθηκα οραματιζόμενη πώς είναι η ζωή των οδηγών, των φορτηγών. Αλλά στο θέμα του Lex Specialis κάνουμε παραπομπή στο Specialis στην οδηγία για την απόσταση των εργαζομένων του 96, η οποία τώρα όμω είναι σε διαδικασία αναθεώρηση και έχουμε μπει σε τριμερεί διαλόγου. άρα κανεί δεν ξέρει ποια θα είναι η έκβασή τη. αφού να σε αναθεώρηση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν. Και αυτό που είπα και εγώ και για τη δική μου τη γνωμοδότηση ακόμα και η ρήτρα της ε, ενσωμάτωσης θα έχει τεράστια τεράστιο αντίκτυπο στη λέξη φεσιάλης. Πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι είναι ε, ευθυγραμμισμένα αυτά μεταξύ τους. Τι είδου συνέπειε δηλαδή θα φέρει η κύρια οδηγία στον ειδικό νόμο, στη λέξη φεσιάλης. Γιατί μερικές φορές κάνουμε παραπομπή σε διάφορους κανόνες αλλά τώρα έχουμε να κάνουμε παραπομπή σε, κανόνα, σε οδηγία του 96 που είναι υπό αναθεώρηση και δεν είμαι βεβαία ότι οι συνάδελφοι των μεταφόρων ξέρουν ότι συζητούμε στους τριμερείς ε, διαλόγους για την αναθεώρηση και κάποιοι κανόνες ίσως να μην ε, ε, προσφέρονται για τον τομέα των μεταφορών. Γι' αυτό και πάντα επιμένω και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των διαφορών θεμάτων. Η κινητικότητα, η απόσπαση των οδηγών που είναι στον τριμερή διάλογο. Όλα αυτά είναι τα θέματα. Βερόνικα λοιπόν, για τη διαμετακόμιση, νομίζω ότι εσύ προς τα εκεί θα τίνεις, αλλά νομίζω και για την ε, απόσπαση και για το θέματα του κυρίου Μπαχ πρέπει να μεριμνήσουμε αυτά όλα να πάνε ε, εκ παραλίλου. Στη δική μου τη γνωμοδότηση σας υπενθυμίζω ότι εγώ έχω συμπεριλάβει από την πρώτη στιγμή την ε, διαμετακόμιση στους κανόνες. Αυτό γιατί υπάρχουν κάποια τα οποία έχουν ε, σαφείς θέσεις αυτό για να εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες για τους οδηγούς. Άρα είναι απαραίτητο τώρα να βρούμε ε, μια καλή ισορροπία για τους οδηγούς γιατί αν υπάρχουν οι κοινωνικές προδιαγραφές προστασίας ας μην είμαστε υπερβολικά περιοριστικοί ως προς τη διάρκεια και, τις, ε, και τα δρομολόγια. Εάν έχουν λυθεί τα θέματα της αμοιβή των οδηγών, χάρη στην απόσπαση, ας μην κινδυνέψει η αγορά των διεθνών μεταφορών. Αυτά λοιπόν. Περιμένω σας δω αύριο να συζητήσουμε στις συνεδρίες των σκιωδών και να προσπαθήσουμε να δούμε συνολικά τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κάρι Γκούε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που μας ε, προσκάλεσε στη συνεδρία των σκιωδών. Ε, θα είναι επικοδομητικές με βέβαια οι επαφές μας. Βεβαίως μπορεί να απέχουμε ως προς τις θέσεις κίνησης σε ορισμένα σημεία, αλλά είμαι βεβαία ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινέ θέσεις για ορισμένα τουλάχιστον για τα ελαφρά φορτηγά όπως και οι σοσιαλδημοκράτες, θέλουμε να περιληφθούν αυτά στην ε, πρόταση. Πρώτα απ' όλα, διότι βλέπουμε ότι το όριο αυτό ε, των ελαφρών φορτηγών το αξιοποιούν ορισμένοι για να ε, καταστρατηγήσουν την νομοθεσία. Ας αποφύγουμε λοιπόν αυτό το κενό. Δεύτερον, καμποτάζ, διαμετακόμιση. Είναι σαφές για μας, υπάρχει καμποτάζ. Και τι είναι, ότι κάνει ένα δρομολόγιο μέσα σε μία χώρα για συγκεκριμένο αριθμό ημερών, κάνει διάφορα δρομολόγια. Εμά εδώ πάνω απ' όλα μα ενδιαφέρουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. ή σε συνθήκε εργασία, ισότιμη αμοιβή για την ίδια δουλειά. Όταν δουλεύει κανεί μέσα σε μία χώρα πρέπει να χαίρει των ίδιων συνθήκων με του εγχώριου εργαζομένου. Πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε το στόχο αυτό, α το συζητήσουμε. Είμαστε ε, διατεθειμένοι να συζητήσουμε. Στόχος μας και πρότασή μας είναι περιορισμός της διάρκειας του καμποτάζ και περίοδος ανάπαυσης, cool off. Δηλαδή μια περίοδος μέσα στην οποία θα γίνεται διαμετακόμιση και μετά μια περίοδος ανάπαυσης ή διακοπής, το cool off, μέσα στην οποία δεν θα μπορεί κανείς να ξανακάνει καμποτάζ. Έτσι ώστε πράγματι να πρόκειται για μια διαμετακόμιση κατ' εξαίρεση και όχι ε, απεριόριστη χρήση αυτής της ευχέρειας. Εμείς προτείνουμε το επταήμερο, αλλά μπορούμε να δεχθούμε διαφορετικά μοντέλα, να στα συζητήσουμε. Το βασικό είναι να γίνει σεβαστή αρχή ότι για ίδια εργασία θα δίδεται ίδια αμοιβή. Η κυρία Ανταλή για τους πράσινους. Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητή Βερόνικα. Το γνωρίζω καλά το θέμα αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητούμε. Ξεκινώντας όμως θέλω να σε ευχαριστήσω για όλη σου τη δουλειά και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημαντικά σημεία αυτής της συζήτηση. Η ίδια μετακόμιση καταρχά είχε θεσπιστεί για να μην γυρνούν άδεια στην έδρα του τα φορτηγά. Δόθηκε λοιπόν αυτή η δυνατότητα την οποία υπερεκμεταλλεύτηκαν και τελικά καταστρατήγησαν ε, σε σχέση με το αρχικό στο χωρισμένο και έτσι προέκυψαν συνθήκες απολύτως αθέμητου ανταγωνισμού και έτσι τώρα είναι επιτακτική η ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί και να περιοριστεί ως εκ τούτου το καμποτάζ. Το καμποτάζ και γι' αυτό κάνω την πρόταση για έναν περιορισμό στην εβδομάδα ε, αυτής της δραστηριότητας. Αντίστοιχα, προτάσεις βλέπουμε στο Συμβούλιο ή προτάσεις σχετικές με τη λεγόμενη συμμαχία του οδηγού και βλέπουμε ότι μπορεί το Κοινοβούλιο να είναι φιλόδοξο στις απαιτήσει του. Η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει σύσσωμη για την αρχή αυτή, γιατί είναι χρόνια που την επιδιώκουμε, ας την συγκεκριμενοποιήσουμε επιτέλους. Και θα ήθελα να περάσω, που το έφερα βέβαια και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, στο θέμα της πλαισίωσης των ελαφρών φορτηγών οχημάτων. Δεν είναι φυσιολογικό να απαλλάσσονται από την υποχρέωση της νομοθεσίας όπως έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Υπάρχουν πολλές μεταφορικές εταιρείες που όλο και περισσότερο ε, χρησιμοποιούν αυτά τα μικρά, τα ελαφρά φορτηγά για να καταστρατηγήσουν την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία με απολύτως αρνητικές συνέπειες και για την προστασία του περιβάλλοντος γιατί αντί για ένα βαρύ όχημα έχουμε δεκάδες ελαφρά φορτηγά που κυκλοφορούν στους δρόμους. Έχουμε θέματα σε σχέση με την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές αλλά και τις συνθήκες εργασίας των οδηγών και γενικά των εργαζομένων του κλάδου. Είναι απαραίτητο λοιπόν επιτακτική ανάγκη να ενσωματωθούν τα ελαφρά φορτηγά στην νομοθεσία. Χαιρετίζω λοιπόν τις τροπολογίες των συναδέλφων και κυρίως των κυρίων Μπαχ και Ροσφόρ που επιδιώκουν αυτό το στόχο. Τελευταία παρατήρηση για τους ελέγχους και τις κυρώσεις, γιατί έχω καταθέσει τροπολογία όπου προτείνω επιχειρήσεις που δεν τηρούν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να περιλαμβάνονται σε μαύρη λίστα αντίστοιχη με αυτή των αεροπορικών μεταφορών γιατί στις αεροπορικές μεταφορές αγαπητοί συνάδελφοι υπάρχουν εταιρείε που έχουν μπει σε μια μαύρη λίστα που ένας πολίτης ε, θα φροντίσει να μην χρησιμοποιήσει γιατί ξέρει ότι δεν ε, ακολουθούν ε, τις διατάξεις νομοθεσίες, ότι δεν είναι ασφαλής. Το ίδιο λοιπόν με, τη, με αυτό που συμβαίνει στι αεροπορικέ μεταφορέ πρέπει να κάνουμε και στι οδικέ. Να μπουν σε μαύρη λίστα αυτέ οι επιχειρήσει εφόσον δεν τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και πρέπει βεβαίως και να απαγορευθούν οι δραστηριότητες διεθνικών μεταφορών. Πρέπει να υπάρχει μια αποπτία βεβαίως παρακολούθηση αλλά και επικαιροποίηση από την Υπηρεσία για την Εργασία που πρόκειται να θεσπιστεί και θέλω επί τη ευκαιρία να χαιρετήσω τις τροπολογίες των συναδέλφων από το ΕΛΚ της Γαλλίας για το θέμα των υπηρεσιών γιατί βρισκόμαστε σε μια κέρια στιγμή, σε ένα σταυροδρόμι για το μέλλον της Ευρώπης, είτε θα δράξουμε την ευκαιρία και θα πούμε ότι κοιτάξτε, επενδύουμε στο ευρωπαϊκό όραμα και θεσπίζουμε αυτή την ευρωπαϊκή υπηρεσία, είτε πολύ γρήγορα, σας διαβεβαιώ, οι ευρωσκεπτικιστές και όσοι θέλουν να καταστρέψουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα θα έχουν αρκετή τροφή για να μας πλήξουν για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαχτά. Από το EFTD δεν υπάρχει άλλος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια. Πραγματικά πάρα πολύ εκτίμησα ε, την ε, πραγματικότητα της προηγούμενης ομιλήτρια όσον αφορά τη, το διπλασιασμό των ελέγχων για το καποτάζ. Το είπα και προηγουμένω. Όταν υπάρχει καμπιτάζ, υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ, ε, υπάρχουν αθέμητε πρακτικέ. Ε, οπότε πρέπει να καταργήσουμε το καμποτάζ. Και κάθε φορά που λέω ότι το καμποτάζ άρχισε να ισχύει για να μην γυρίζουν άδεια τα φορτικά, μα όταν μιλάμε για διαθέσει μεταφορές οδικές, ε, ποτέ δεν γυρίζει κανείς πίσω άδειος, περνάει από χώρες, πολλές χώρες και ε, υπάρχει τρόπος να γίνουν προτάσεις ε, που να επιτρέπουν ε, να γίνει μια μεταφορά από μία χώρα σε μια άλλη χώρα. Οπότε είναι, το επιχείρημα είναι εντελώ λανθασμένο. Όσον αφορά το καμποτάζ, αν το καταργήσουμε θα πάνε όλα πολύ καλύτερα ή αν διατηρήσουμε τον καποτάζ πρέπει οι οδικές μεταφορές να παραμείνουν ε, στο πεδίο εφαρμογής ε, της τροποποιημένης οδηγίας ε, περί απόσπασης εργαζομένων. Κυρία ε, Λαμπάνιοβα, πώς θα το υπολογίσετε αυτό, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Αν περνάει ένας οδηγός μία μέρα στη Γερμανία με τις συνθήκες που ισχύουν εκεί, μετά πάει στο Βέλγιο για ένα πρωινό, ένα πρωινό για τις συνθήκες της Βελγικές, μετά στη Γαλλία, ισχύουν οι γαλλικές συνθήκες, ε, τι να κάνουμε τώρα, είναι ένα... ε, ε, ε δύσκολο θέμα ε, και λέτε απλώς ότι το επιχείρημα είναι να μην γυρίσει πίσω άδειο ένας, ε, ένας οδηγός. Ε, μα κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει κατάχρηση, αλλά αυτό είναι, γίνεται επίτηδες. Πρέπει σε, όλες τις, σε όλους τους κανόνες, σε όλες τις υποχρεώσεις να αναφέρεται αυτό το κομμάτι που αφορά το καμποτάζ. Ευχαριστώ πολύ. Ντανούτα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και εγώ επιθυμώ στην Επιτροπή μας να καταλήξουμε σε ένα καλό έγγραφο και το λέω αυτό απευθυνόμενοι κυρίως ε, στους συγητές οι οποίοι ασχολούνται με, το, με την πολύ περίπλοκη δέσμη μέτρων για την ε, κινητικότητα. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει έλλειψη οδηγών ε, και αυτό δεν αφορά μόνο τη Δυτική αλλά και την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε προτεραιότητα να δημιουργήσουμε καλές συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς για να έχουν ικανοποιητικό χρόνο Λοιπόν Οδήγηση και ανάπαυσης και βεβαίως πρέπει να υπάρχουν και εξασφαλίσεις για την οδική ασφάλεια για να διασφαλιστούν όλα αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτά που λέει ο κύριος Ζορζ Μπαχ στους ε, χρόνους οδήγησης ε, και ανάπαυσης. Για να επιτύχουμε την ε, απαραίτητη ευελιξία πρέπει να πλουστευτούν οι κανόνες για τους χρόνους ανάπευσης. Δεν είναι δυνατόν οι κανόνες ε, να διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα και οι οδηγοί να διατρέχουν κίνδυνο να τους επιβληθούν πρόστιμα. Ε, θα πρέπει το χρόνο να τον επικίνουμε από δύο σε τέσσερις εβδομάδες. Ίσως οι οδηγοί να μπορούν να έχουν χρόνο ανάπαυσης ακόμα και πέντε ημέρες. Αυτό είναι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον και ε, με συγχωρείτε προς την οικογένεια και γι' αυτό ε, καταθέσαμε και σχετική πρόταση. Όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Μπαχ, θεωρώ ότι πρέπει να ρυθμίσουμε και το θέμα του χρόνου ανάπαυσης ε, στην καμπίνα οδηγού τα κράτη-μέλη πρέπει να επενδύσουν σε φυλασσόμενους ε, χώρους στάθμευσης. Πολύ σημαντικό αυτό, το είπε και ο κύριος Μπαχ, γιατί δεν είναι δυνατόν ο οδηγός την ώρα που κοιμάται να είναι και υπεύθυνο για την ε, φύλαξη των εμπορευμάτων. Σήμερα, από ό,τι φαίνεται, ε, τα εμπορεύματα όμως είναι ασφαλή μόνο αν είναι ο οδηγός παρόν. Και μόνο έτσι ασφαλίζονται τα εμπορεύματα οποτεδήποτε μεταφέρονται στο εξωτερικό. Στην καμπίνα του οδηγού να μπορεί να επιτρέπεται χρόνος ανάπαυσης μόνο και εφόσον η καμπίνα είναι σωστά εξοπλισμένη. Ε, πριν από μερικά χρόνια είχαμε ρυθμίσει το θέμα αυτό έτσι ώστε να υπάρχουν και ικανοποιητικές ρυθμίσεις για τους οδηγούς. Αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται αν δεν υπάρχουν ε, αρκετοί ε, χώροι φυλασσόμενων πάρκινγκ. Νομίζω ότι όλα αυτά αποτελούν και κίνητρο για τα κράτη μελη Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να ελέγχει την κατάσταση και να ενταρρύνει τα κράτη-μέλη να σημειώσουν πρόοδο. Όσον αφορά τώρα την ε, πρόταση της ε, κυρίας ε, Λόπε Φοντανιέ. Εδώ θα ήθελα να αφαιρθώ λιγάκι στο θέμα που αφορά στις ενδομεταφορές στο καμποτάζ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον, χρειάζεται τις ενδομεταφορές και γι' αυτό πρέπει να απελευθερωθεί ο τομέας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απελευθερώσει λιγάκι τον περισμένο αριθμό των ενδομεταφορών η Κάριν πολύ σωστά επισήμανε ότι οι ενδομεταφορές θα πρέπει να έρχονται κατά το ανώτερο σε 7 ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Έφαγε, έφυγε κρίμα είναι. Δεν είναι τυχαίο που έβαλα σήμερα ένα πράσινο ρούχο. Ε, γιατί νομίζω ότι συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με την Καρίμα Ντελή και με άλλου συναδέλφου για το θέμα αυτό, αλλά σοβαρά τώρα. Μία ακόμη φορά δεν έχω αιμονία, απλά είναι ένα ζήτημα που το δουλεύω εδώ και πολλούς μήνες, ε, το θέμα των ελαφρών οχημάτων που ε, είναι εκτός κάθε νομοθεσία. Γιατί? γιατί είναι ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε. Ακούω αυτούς που μου λένε όπως ε, η, Μαρτίν, η, η, η Μαρτίνα ότι δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία για τα ελαφρά οχήματα και ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει και συνεπώς δεν χρειάζεται να νομοθετήσουμε. Μα κοιτάξτε, επειδή δεν υπάρχει αλλαγνώριση νομική, είναι δύσκολο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα. Άλλοι μου λένε ότι είναι ένα πρόβλημα που είναι δευτερεύον, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει νομοθεσία, νομοθεσία γι' αυτό. Αντιθέτω, ο, ω νομοθέτε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επέμβουμε όταν τα προβλήματα είναι δευτερεύοντα από το να ε, υπάρξει μια εκθετική αύξηση του φαινομένου και να είναι τότε πάρα πολύ δύσκολο και δεν θα μπορούμε να πάμε προ τα πίσω. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για κάθε ένα από τα ε, ζητήματα να μπορούμε να πάμε προ την κατεύθυνση ενσωμάτωση ε, στην νομοθεσία και στους ευρωπαϊκούς κανόνες ε, την προβληματική αυτή των ε, ελαφρών οχημάτων, να πούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα ε, και όταν σε 3-4 χρόνια ε, θα πούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι μη διαχειρίσιμο, δεν θα βρεθούμε σε μια θέση που να μην έχουμε κάνει τίποτε και να μην μπορούμε πια να πάμε προ τα ε, πίσω. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει πραγματική συνειδητοποίηση του προβλήματο και πρέπει να υπάρξει μια συνένεση και εδώ και στην Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Είμαι από την Γενική Διεύθυνση MOVE. Θα ήθελα να φερθώ σε δύο θέματα, στις ε, δύο προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Lex Specialis, είναι το ένα, και το δεύτερο αφορά χρόνους ανάπευσης και χρόνους οδήγησης και θέμα ταχογράφων. Ο συνάδελφός μου θα σχολιάσει το τελευταίο θέμα που μόλις τώρα συζητήθηκε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι, να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει νομοθετικές προτάσεις ως μία δέσμη μέτρων και λύσεων. Γιατί εμείς ε, είχαμε μία μακρά διαδικασία ε, και ε, ασχοληθήκαμε με όλες τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των οδικών μεταφορών. Τα προβλήματα είναι άρρηκτα συνδεμένα μεταξύ τους, όπως ανέφερε σήμερα και η κυρία Λαμπάγεβα. Ως εκ τούτου, ε, θέματα ανταγωνισμού συζητούνται από κοινού με τις οδικές ασφάλειες και είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει αυτή η προσέγγιση στην αναζήτηση συμβαστικών λύσεων. Δηλαδή, να θεωρούνται όλα αυτά ως μία δέσμη μέτρων. Όσον αφορά το Lex Specialis, προφανώς η διαχωριστική γραμμή είναι το πεδίο εφαρμογής αυτού του ειδικού νόμου. Πρέπει να γίνει κατανοητός ο στόχος ότι πρέπει να υπάρχουν, υπάρχει η σωστή συνεπής ε, εφαρμογή ε, των κανόνων περί απόσπασης εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών, χωρίς διοικητικό φόρτο. Ε, υπόθηκε ότι η Κομισιόν επιφέρει χάος, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι η πρόταση Κομισιόν είναι η απάντηση, στην κατάσταση που υπάρχει τώρα, όπου έχουμε διάφορα διοικητικά μέτρα και όπου τα διάφορα κράτη-μέλη εφαρμόζουν διαφορετικές διοικητικές ηχητικές ρυθμίσεις. Το ένα κράτος μέλος θέλει δήλωση με φάξ, το άλλο με ηλεκτρονικό μήνυμα, το άλλο πάλι ε, να καταβάλλεται κάποιο τέλος. Ε, ένα κράτος μέλος θέλει η οδηγία να καλύπτει 6 μήνες, άλλο κράτος μέλος θέλει για κάθε μετακίνηση και μια οδηγία. Εμείς λοιπόν θέλουμε να υπάρχει ένας κατάλογος εναρμονισμένων διοικητικών διατάξεων. Όσον αφορά τώρα το ε, ανώτατο όριο, θέλω να πω ότι εκτός από το ότι προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία. Να ισορροπήσουμε, να εξισορροπήσουμε την προστασία κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και διοικητικέ απαιτήσει για να συνεχίσουν να προσφέρονται υπηρεσίε. Αυτή η ισορροπία ε, προφανώ γίνεται διαφορετικά κατανοητή από εμά ή από εσά. Υπάρχει διαφορετική ερμηνεία. Υπάρχει όμω ένα στοιχείο που πρέπει να έχουμε κατά νου ε, όσον αφορά το κατόφλι, τους κινδύνους και αυτό αφορά και την ε, ε, μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου αν είναι πολύ χαμηλό το ανώτατο όριο τότε προκύπτουν κίνδυνοι ε, αυτό μπορεί να προκαλέσει και την εκπεριτροπή απασχόληση των εργαζομένων των οδηγών για να παρακαμφθεί ο κανόνας τι είναι η λύση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, τη δική μας την πρόταση για χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι υποστηρίζεται μια νέα πρόταση για την επιστροφή στο σπίτι. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές λύσεις, αλλά όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όπως εμείς ερμηνεύουμε τις τροπολογίες, ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει αρκετός χρόνος ανάπαυσης για τους οδηγούς και για την υγεία τους και για την οδική ασφάλεια. Υπάρχουν βέβαια κάποια νέα στοιχεία τα οποία εμεί έχουμε καταγράψει και έχουν προκύψει από τις τροπολογίες. Καταρχήν όσον αφορά η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συστήσει αυτή την αρχή, την ΕΛΑ, η οποία θα ασχολείται με θέματα εφαρμογής και διοικητική συνεργασία στον τομέα των οδικών μεταφορών. Αυτές οι τροπολογίες λοιπόν που έχουν κατατεθεί είναι πολύ επίκαιρε γιατί βαδίζουν ε, με αυτά που ε, προτείνουμε και εμείς. Τώρα, ασφαλής ε, χώρη στάθμευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Χάρη της βοήθειας από τον ε, προϋπολογισμό, από τα κονδύλια που διατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα μπορούμε πλέον να εφαρμόσουμε μία μελέτη για τις δυνατότητες που υπάρχουν έτσι ώστε να προκύψουν τέτοιοι ασφαλείς χώροι στάθμευσης. Κατόπιν, όσον αφορά τα LCVs ε, γνωρίζετε ε, ότι όσον αφορά τα ελαφρά οχήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για να υπάρχει επαγγελματισμό στον τομέα. Ε, Βεβαίω για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα υπάρχει πρόταση να εγκατασταθούν σε αυτά ταχογράφη. Ε, αυτό όμως αφού προηγηθεί μια ανάλυση κόστους ωφέλους για τον τομέα. Και ως προς τους ταχογράφους η εισαγωγή των εφιών ταχογράφων άκουσα ότι το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προβλέπει το 2030 ως καταληκτική ημερομηνία για να έχουν εξοπλιστεί όλα τα οχήματα με ευφυείς ταχογράφους. Δεν το είπαμε εμείς αυτό. Ε, εμείς ε, δεν προτείναμε αλλαγή της μεταβατικής περίοδου το 2014 εγκρίθηκε μεταβατική περίοδος από τους νομοθέτες. Πάντως εμείς έχουμε αναθέσει μία μελέτη ε, για να ε, αναλυθούν, ε, να λυθεί το κόστος και το όφελος της εκ των υστέρων και της αναδρομικής εγκατάστασης των ταχογράφων. Θα προκύψουν λοιπόν στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν την έγκαιρη εγκατάσταση των ταχογράφων. Και τέλος θέλω να πω ότι αν μιλάμε για την εγκυρή εγκατάσταση των ταχογράφων θα πρέπει να ε, δούμε και το ότι θα πρέπει να υπάρχουν και εποπτικές αρχές ε, με ένα μηχανισμό εντοπισμού εξ αποστάσεως. Αυτές οι αρμόδιες αρχές να έχουν αυτόν τον εξοπλισμό γιατί αλλιώς οι ταχογράφοι είναι άχρηστοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φοντανιέ για το σχέδιο γνωμοδότησής της ε, υπάρχουν μερικές ιδέες ε, που τις βλέπουμε θετικά και που μας βρίσκουν σύμφωνους, όπως ε, για παράδειγμα η εστίαση, ως, ε, η της επιβολής των διατάξεων περί καμποτάζ. Είναι επίσης ένας στόχος τον οποίο συμμερίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να είναι οι σχετικοί κανόνες σαφείς, απλοί, αλλά πρέπει να γίνεται και έλεγχός του στην πράξη. Υπάρχει συνεπώς ανάγκη ε, Σωστή επιλογή των κανόνων. Όσον αφορά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, έχουν υποθεί ήδη αρκετά. Θα ήθελα απλώς να σημειώσω ότι πράγματι προσπαθήσαμε να έχουμε μια εξισορροπημένη προσέγγιση αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των οχημάτων αυτών και ότι χρησιμοποιούνται και στην διεθνή κυκλοφορία. Πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις ως επιτοπλίστων ε, και θα έπρεπε να αποφύγουμε την υπερβολική ρύθμιση. Ε, ωστόσο βλέπουμε την ανάγκη να δράσουμε τώρα γιατί όπως ήδη υπόθηκε αν δεν κάνουμε τίποτε για τέτοιου είδους ε, μεταφορές τώρα στην επόμενη αναθεώρηση σε 10-15 χρόνια ε, το φαινόμενο μπορεί να έχει ενταθεί πολύ περισσότερο. Είναι λοιπόν ενδιαφέρουσα ιδέα το να επικεντρωθούμε στις μεταφορές επαγγελματικών οχημάτων που έχουν πραγματικό διασυνοριακό αντίκτυπο ε, και στους διεθνείς ε, μεταφορές, στους διεθνείς μεταφορείς που είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περισσότερο κάτι για το άρθρο 3 παράγραφος 2 του, 1071, δηλαδή, του κανονισμού 1071, δηλαδή τη δυνατότητα επιπλέον κριτηρίων από πλευρά κρατών μελών ε, για τα επαγγέλματα εκτός από αυτούς που αναφέρονται στον κανονισμό. Η προσέγγιση μας είναι ότι χρειαζόμαστε κανόνες που να είναι κοινοί. Χρειαζόμαστε περαιτέρω εναρμόνιση. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να έχουμε ένα ευρύτερο σύνολο ε, κριτηρίων ε, υπό τους κανόνες εγκατάστασης, όμως δεν θα θέλαμε να ε, εξαλείψουμε αυτήν την, θα θέλαμε μάλλον να εξαλείψουμε την δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή μονομερός να επιβάλλουν κάποιους κανόνες ε, ε, στους οδηγούς τους και στις οδικές μεταφορές. Ένα ακόμη πολύ ευαίσθητο ζήτημα είναι αυτό του καμποτάζ Πράγματι, εμείς θεωρούμε ότι είναι ένας καλός συμβιβασμός η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ μιας αποτελεσματικής αγοράς, απλών κανόνων που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, αλλά παράλληλα βλέπουμε ότι η κατάσταση σήμερα, και έχει αναφερθεί αυτό πολλές φορές ε, σήμερα, ε, η εθνική μεταφορής ε, σε μερικά κράτη-μέλη βρίσκονται υποπίεση ανταγωνισμού από ξένους μεταφορείς, ακόμη και αν ο μακροπρόθεσμος ε, στόχος μας είναι να έχουμε μία ενιαία αγορά οδικών ε, μεταφορών. Δεν έχουμε φτάσει εκεί σήμερα και δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα προς την απελευθέρωση και την, το άνοιγμα ε, των αγορών. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, Βερόνικα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ στο μια και θα συναντηθούμε αύριο. Μερικές παρατηρήσεις. Πρώτον, ηλεκτρονικό μητρό ή ηλεκτρονικά μητρό, εθνικά. Όπου το έχουμε στο κείμενο. Έχουμε καταθέσει συμβαστική τροπολογία καθώς ε, στην ε, Επιτροπή μιλούσαμε για τον κανονισμό, για το ενεργητικό, του ε, όγκου των συναλλαγών κτλ. Καταθέσαμε λοιπόν μια συμβαστική τροπολογία που πιστεύω αύριο μπορούμε να συζητήσουμε ενδελεχέστερα για να δούμε τι άλλο θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Δεν πρόκειται για κατάργηση λοιπόν, αλλά για τροποποίηση. κανόνε που ισχύουν για του αποσπασμένου εργαζομένου. Συμφωνώ ότι πρέπει να καλύπτονται σε ένα κείμενο, Μαρτίνα, και δει τη γνωμοδότηση τη δική σου. Για τη διαμετακόμιση, καμποτάζ που είναι το πιο περίπλοκο θέμα, θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και συμφωνούμε πιστεύω να υπάρχουν και οι έλεγχοι και η εγγύηση του, ε, της επιστροφής της αιστείας ούτως υπήν. Δεν μπορούμε βεβαίω και να καταστρέψουμε την εσωτερική αγορά, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε την τήρηση των κανόνων. Μπορούμε σε αυτό να συμφωνήσουμε νομίζω συζήτηση υπάρχει, αρκετό περιθώριο για συζήτηση δηλαδή, και τι είναι αρκετά περίπλοκα τα θέματα. Είμαι βέβαια ότι οι συζητήσεις ε, θα είναι και αλλά και πολύ ενδιαφέρουσε. Και προσβλέπω σε μια θετική έκβαση και ω προ τα ελαφρά φορτηγά. Περίπλοκο επίση θέμα. Γι' αυτό είχα κάνει δεκτή την πρόταση του Ζοσμπαχ. Μπαχ. Ενδιαφέρουσα μου φάνηκε και θεωρώ ότι πρέπει να τη συζητήσουμε όχι 3,5 τόνους και κάτω αλλά το, η ουσία είναι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Μια καλή λύση λοιπόν, ε, αυτά από μένα και βεβαίως βεβαίως θα λάβουμε υπόψη και την γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής των Μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ε, πρακτικά μόνο, όχι για το περιεχομένο, για ένα τόσο σημαντικό νομοθετικό θέμα θα έπρεπε να είμαστε καλύτερα εκπροσωπούμενοι εδώ. Δεν νομίζω ότι ήταν ε, συνετό το ότι μπήκε στην ημερήσια διάταξη Δευτέρα απόγευμα στις 3 πρώτο θέμα, γιατί κάποιοι δυσκολεύονται να φτάσουν στην ώρα του στη συνεδρίαση. Έπρεπε να έχουμε περισσότερο χρόνο για μεγαλύτερη προσέλευση. Και επίση την Πέμπτη μόλι άλλαξε η ημερήσια διάταξη. Δηλαδή, αν κάποιο είχε ανηλυμένε υποχρεώσει, εγώ είχα άλλη επιτροπή, μάλιστα έπρεπε να πάω από εκεί, μετά να έρθω εδώ. Και ω εισηγήτρια ακόμη δεν είχα νωρίτερα ενημερωθεί από ε, για την αλλαγή αυτή τελευταία στιγμή έραβα γνώση. Παρακαλώ λοιπόν σε τέτοια νομοθετικά θέματα που δεν είναι πολλά στις αρμοδιότητες μας να είμαστε σε επαγρύπνηση. Αυτό ως σύσταση για ε, κάποια επόμενη ευκαιρία. Ο πρόεδρος βεβαίως πρέπει να επαγρυπνούμε σε αυτά τα θέματα. Ειδικά στα σημαντικά νομοθετικά. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα. 27 ή 28 Μαρτίου για την Επιτροπή, 24 Μαΐου για την Τράνα και δεν ξέρω εάν αντί να μετράμε πρόβατα για να κοιμηθούμε θα μετράμε φορτηγά αλλά αύριο να είμαστε όλοι ε, σε επαγρύπνηση και να προλάβουμε έχουμε ψηφοφορίες, μιλούμε για τις μεταφορές υπάρχει και απεργιακή κοινοτοποίηση αύριο στις Βρυξέλλες που αφορά και τους σιδηροδρόμους αλλά και τα τραμ, τα μετρό, τα λεωφορεία να προλάβετε λοιπόν και να μην σας πιάσουν στον ύπνο. Αύριο λοιπόν. Και τα ξαναλέμε με τις ψηφοφορίες αύριο. Ευχαριστώ.